morning, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει η πρόεδρος, γιατί προεδρεύω, γιατί η Ντόρις Πάκ πρέπει να πάει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να μιλήσει για την έκθεσή της για τη Βοσνία και γι' αυτό προεδρεύω στη θέση της στις 10 πρέπει να πάω σε μια συνάντηση συντονιστών. Αν έχει γυρίσει η Ντόρις θα προεδρεύσει αυτή, αλλιώς κάποιος από τους συναδέλφους αντιπροέδρους. Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα έχουμε την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Έχετε σχόλια ή παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις ή ενστάσεις. Όχι. Ωραία. Δεύτερο σημείο. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου. Έχετε στο φάκελό σας τα πρακτικά. Όσοι ήθιστε, εάν δεν εγερθεί κάποια αντίρρηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας, θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Ευχαριστώ. Τρία. Ανακοινώσεις Προέδρου. Διερμηνευτικές διευκολύνσεις. Όλες τις γλώσσες εκτός από τσεχικά, εστονικά, λιθουανικά, λετονικά, μαλτέζικα και σουηδικά. Και πάμε στην, στις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με τον εξυγχρονισμό του συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, η έκθεση Τσέκες και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσέκες αν θέλει να λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη τιμή ήταν να έχω αυτή την έκθεση καταφέραμε να έχουμε με όλες τις πολιτικές ομάδες και τους κοιόδης εισηγητές μια πολύ καλή συνεργασία και θέλω να τους ευχαριστήσω. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ντιβιντάλοβα, τον Λουίτζι Μπερλίνγκουερ, τον Ζαν Γκάλσκι, τον Αραμπατούν. και τον κύριο Λορέντζο και είχαμε και σημαντική υποστήριξη από τις ε, διάφορες ε, από τη Γραμματεία της Επιτροπής μας, από την Επιτροπή των ε, Περιφερειών, από την Ένωση Πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί έχουν υποστηρίξει την έκθεση αυτή και θέλω να σας ευχαριστήσω. Thank you, Mr. Turkish, Mrs. Η κυρία Νεβετάλοβα θέλει να λάβει το λόγο. Ένα μικρό αίτημα. Θέλουμε να αλλάξουμε τη σειρά της ψηφοφορίας. Θέλουμε να αλλάξουμε τη σειρά των τροπολογιών 8 και 34. Νομίζω ότι 34 είναι γενικότερα της 8. Θα ήθελα να ψηφιστεί πρώτα η 34 και μετά η 8. Ο εισηγητής έχει συμφωνήσει. Θα ήθελα πρώτα να σας ζητήσω να γίνει έτσι. Okay. Συμφωνείτε? Θα πράξουμε όπως συζητήσατε. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. <clears throat> Παράγραφος 1, τροπολογία 28. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 29. Ψήφι. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Η 30 εξέπεσε. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ και εδώ Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 ο εισηγητής κατά ψήφι υπέρ. Ας το κάνουμε ηλεκτρονικά, είναι πιο εύκολο. Πάρτε τις κάρτες σας παρακαλώ. Δεν έχετε κάρτα. Okay, then we have to count you. Θα σας μετρήσουμε πάντως. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Okay, we close the vote. τις ψηφοφορίες. 12 υπέρ, 12 κατά μία αποχή απορρίπτεται κατά συνέπεια. Α, συγγνώμη. Και οι δύο ψήφοι θετικές χωρίς κάρτα. Εντάξει, τότε εγκρίνεται. Συγγνώμη. Α, εντάξει, είναι μία ακόμα ψήφος υπέρ, μία ψήφος κατά, οπότε απορρίπτεται. Λείπαμε πολύ. Απορρίπτεται. 33 ο εισηγητής κατά ψήφι υπέρ αυτή ήταν η υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην παράγραφο 1α τροπολογία 34 η 34 πρώτα ο εισηγητής κατά ψήφι υπέρ Α, ηλεκτρονικά καλύτερα γιατί δεν είναι εύκολο έτσι. We the vote. Πέρας. 12, in favor, 12 υπέρ 14 κατά απορρίπτεται. Πηγαίνουμε τώρα στην 35 λέει η πρόεδρος. Συγητής κατά ποιο ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεν ψηφίσαμε την 8 Ναι, ναι, συγγνώμη. Γυρίσουμε ένα βήμα πίσω για να ψηφίσουμε την τροπολογία 8. Το γυναικών εισηγητής είναι κατά ψήφι υπέρ. κατά αποχές απορρίφθηκε παράγραφος 2 συμβιβαστική 1 ο εισηγητής είναι υπέρ προφανώς ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην παράγραφο 2α, τροπολογία 42, Ο εισηγητής είναι θετικός, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2α παράγραφος 43 ψήφι ε, υπέρ, ο συγκεκριτής είναι κατά αποχές εγκρίνεται. 44 θετικός ο συγκητή, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, παράγραφος 45, αρνητικός ο εισηγητής, Ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 θετικός ο εισηγητής. <clears throat> Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 <clears throat> θετικός ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 48 θετικός εισηγητής ψήφι υπέρ ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας 15 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 449 αρνητικός ο εισηγητής ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 πάλι αρνητικός ο εισηγητής ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ ο εισηγητής, ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, εγκρίνεται, εγκρίνεται, εγκρίνεται λέω. Συγγνώμη. Δεν θέλω να αλλάξετε τον τρόπο που κάνετε ψηφοφορία, αλλά μπερδευόμαστε με αυτά που λέτε για τον εισηγητή. <clears throat> Μπορούμε να λέμε απλώς υπέρ κατά ε, αποχές με το να λέτε ποια είναι η σύσταση του εισηγητή κάθε φορά μπερδευόμαστε. Εντάξει, δεν θα λέω τίποτα για τον εισηγητή, το έχετε στην, στον κατάλογό σας. 52 υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονικά θα το κάνουμε αυτό. 52 ηλεκτρονικά. Άρχεται. 15 υπέρ 11 κατά 2 αποχές Κρίνεται. Παράγραφος 5 τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ υπέρ είπα εντάξει 65, 65. Ψηφίζουμε την 65. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ ηλεκτρονικά για την 68 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 14-14 απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 με προφορική τροποποίηση 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ ηλεκτρονικά 112 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 14 με 15 απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές <clears throat> απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος εντάξει 119 1-1-9 We close Πέρας της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 κατά πίπτη, 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά,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 ε, απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 αποσύρεται 134 υπέρ να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση ποιος είναι υπέρ της 134 Πέραση της ψηφοφορίας. 15 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Να κάνουμε έναν έλεγχο για την 135. Πέραση της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 136 υπέρ. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 139 υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. 17 υπέρ. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. να γίνει έλεγχος παρακαλώ 18 υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. 143 υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση και πάλι. Αλλάζουν συνέχεια οι πλειοψηφίες. 15 υπέρ, 13 κατά εγκρίνεται. 144 υπέρ. Υπέρ για την 144 κατά. Απορρίπτεται η πλειοψηφία είναι κατά. 145. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά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 αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τώρα 157 υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. 157. 15 υπέρ, 14 κατά εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 171. 14 υπέρ, 14 κατά, απορρίπτεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ Δεκαεπτά υπέρ, 10 κατά εγκρίνεται, 177 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ συγγνώμη κατά τμήματα για το πρώτο τμήμα υπέρ ηλεκτρονικός. Πρώτο τμήμα της 180. 13, υπέρ, 14 κατά απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, καλύτερα είναι να... Α, όχι. Για το δεύτερο τμήμα λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 8 16 υπέρ, 12 κατά εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, δύσκολο να ελέγξουμε. 16 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ επαλήθευση Δεκαπέντε 15 υπέρ 11 κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, να κάνουμε μια επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 20. «13 υπέρ, 14 κατά, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προχωρούμε στην 22, κατά τμήματα, υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά, δεύτερο τμήμα για την 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23, υπέρ. Επαλήθευση για την 23. 11-18 απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 226 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική 3 και επιτροπολογία 4 υπέρ, επαλήθευση. Ο 20. Συγγνώμη, 21-7 εκρίνεται βεβαίως. Και 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών. Suggestion A. Who's in favor? Για την A. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. B. Υπέρ. Να κάνω μια επαλήθευση. Δώδεκα, δεκαεπτά, απορρίπτεται. C. Υπέρ. Επαλήθευση. Δεκατέσσερα, δεκαπέντε. Απορρίπτεται. D. Να κάνουμε μια επαληθευση δεκατέσσερα δεκαπέντε, απορρίπτεται ή e ίδια πλειοψηφία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. F υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά επαλήθευση Fourteen to fourteen. 14, 14 απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχέ απορρίπτεται. 16. 16 υπέρ, κατά, επαλήθευση. Γιατί 16.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 11-16 απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ωραία. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ. «25 ψήφι υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές». Συγχαρητήρια κύριε Τσέκης. Ωραία. Περνάμε στην ε, έκθεση Lockerguard. Δυστυχώ ο κύριος Lockerguard δεν είναι μαζί μα σήμερα. Θέλει κάποιο άλλο να λάβει το λόγο από την ομάδα φιλελεύθερων. Ναι, εγώ. Βρίσκεται στην Νότια Αφρική ο κύριος Λόκεγκάρτ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στείλει μια αποστολή εκεί ε, είναι ο κ. Λόκεγκαρντ με την κυρία Βερχόγεν. Ε, τίποτα. Θα, να ευχηθεί απλώς ε, καλή ψηφοφορία, θέλω ο κ. Λόκεγκαρντ ε, μέσω μου. Sorry. Um, we start with... Ωραία. Ξεκινάμε την τροπολογία 1, παράγραφος 2. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. «11 υπέρ 18 κατά απορρίπτεται». Τροπολογία 4 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Περνάμε στην έκθεση... Okay, we come to the by Mrs. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Βερζιά. Θέλετε το λόγο κυρία Βερζιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιοδησηγητές και το προσωπικό των ομάδων καθώς επίσης και της Γραμματείας του Ευρωκοινοβουλίου ότι οργανώσαμε αρκετές συνεδριάσεις για αυτή την νομοθετική γνωμοδότηση. Ομολογώ ότι ήταν η πρώτη φορά για μένα, ε, πρώτη φορά που χρειάστηκε να συντάξω μια τέτοια νομοθετική νομοδότηση. Ε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για μένα, ιδιαίτερα δεδομένου του θέματος. Ε, με ξέπληξε η συζήτηση με τους σκιώδης ηγητές ξαφνικά εμφανίστηκαν χτες ε, αντιρρήσεις οι οποίες δεν είχαν εκφραστεί στις συνεδρίαση μας. Ε, θα προσπαθήσω να υποβάλω ενδεχομένω κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίες. Εγώ προσπάθησα να συμπεριλάβω όλες τις, εκφράσεις, όλες που είχαν εκφραστεί, ξαφνικά όμως εμφανίστηκαν αντιρρήσεις χτες. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Ξεκινάμε τις υποφορίες. Ο κ. Yeah, ε, πληροφοριακά να σας πω το εξής, να ρωτήσω. Γιατί η τελική ψηφοφορία δεν έγινε ηλεκτρονικά στην προηγούμενη, στην προηγούμενη γνωμοδότηση του κ. Λόκεγκάρτ. Γιατί δεν έγινε ηλεκτρονικά η τελική ψηφοφορία. Θέλετε να γίνει ηλεκτρονικά, λέει η πρόεδρος. Υπάρχει λόγος που δεν έγινε ηλεκτρονικά. Ήταν σαφής η πλειοψηφία, αλλά αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Πάντοτε υπάρχουν, πάντοτε στις τελικές ψηφοφορίες, ε, σχεδόν πάντοτε, οι ψηφοφορίες ε, είναι σαφείς, οι πλειοψηφίες είναι σαφείς στην τελική ψηφοφορία. Ε, γι' αυτό ρωτάω. Αν προτείνετε να την κάνουμε ηλεκτρονικά, κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρχε κανένα είδου ιστεροβουλία. Ωραία. Κάνουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την τελική εφορία της έκθεσης Locking Okay. Okay. Ωραία, 25 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Ωραία. Επιστρέφουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Βερζιά. Ξεκινάμε με την τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ ηλεκτρονικά παρακαλώ Δεκαεπτά υπέρ 11 κατά εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. Ωραία, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 56. Oh, 11 18, υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται. Οπότε πάμε στην 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχέται. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Έχει αποσυρθεί. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ 67 λέω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά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 Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 38. ...17 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται... ...39 υπέρ... ...κατά αποχές... ...εγκρίνεται 40 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...13 υπέρ... ...κατά αποχές... ...εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Στη 15 έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Ψηφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πρώτο τμήμα. Τη 44. 16 υπέρ 13 κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 46 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται 47 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται 48 κατά απόχέ. εγκρι... ε, απορρίπτεται 17 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται 49 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται 72 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 και 74 έχουν αποσυρθεί. Περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. ...26 υπέρ, 3 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Βερζιά. Okay, Εντάξει. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Έκθεση Μπένα Ραμπατού. Μαλίκα, θες να λάβεις το λόγο. Απλώς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν συμβάλει στην, ε, ε, στη βελτίωση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ωραία, θα ψηφίσουμε τότε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 2. «11-16 απορρίπτεται». Τροπολογία προφορική 1 στην τροπολογία 3 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Κρίνεται, συγγνώμη, λέει η πρόεδρο. Ναι, ναι. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Έλεγχο στη 5. 13. δεκατρία απορρίπτεται. 6. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 3 συμβιβαστική 1 ψήφι υπέρ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 16-11 εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε, ελέγχουμε, ελέγχουμε 39 11-15 περίφθη. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά από εντάξει θα ελέγξουμε 42 ηλεκτρονικά 11-15 απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα. 23-2, καμία αποχή, συγχαρτήρια στην Μαλίκα. Τελείωσε ο κατάλογος ψηφοφοριών για σήμερα. Πρέπει να φύγω για την Επιτροπή προπολογισμών. Ο κύριο Μπίσκι λοιπόν πρέπει να αναλάβει. Καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έπρεπε να παρουσιάσω την έκθεσή μου για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, γιατί είμαι μόνιμη εισηγήτρια για τα θέματα αυτά. Δεν μπορούσα να είμαι εδώ το πρωί. Χαίρομαι που είναι δίπλα μου ο συνάδελφος Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ ο οποίο θα μα παρουσιάσει τα θέματα του ευρωπαϊκού οίκου ιστορίας ή του οίκου ευρωπαϊκής ιστορία η πρωτοβουλία από τον κύριο Πέτρινγκ, τον πρώην πρόεδρο του οικου Ευρωπαϊκή Ιστορία καλυτερα ξεκινησε αυτη η Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που προετοιμάζει αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο για τον οίκο αυτό παρουσιάστηκε το 2008, το Δεκέμβριο ήδη ενώπιον της Επιτροπής μας και ο χρόνος έχει περάσει, θέλουμε να δούμε πόσο έχει προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Και κύριε Πρόεδρε Ματίνες, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ντόρις. Θα μιλήσω ισπανικά. Μεταξύ άλλων, διότι ως αντιπρόεδρος είμαι και υπεύθυνος για θέματα πολυγλωσσίας, επομένως για λόγους συνέπειας μιλώ πάντα την ε, μητρική μου γλώσσα και θα, αυτό θα κάνω και σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση να έρθω εδώ. Ντόρις, είναι η πέμπτη φορά που έρχομαι. Πέμπτη φορά έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας. Και όπως και να έχει, η κυρία Πακ και η κυρία Παλιαδέλη, η οποία δεν είναι εδώ σήμερα, είναι ιδιαίτερα δραστήριο μέρος της Επιτροπής και συμμετέχουν στην ε, πραγματικότητα και στο Συμβούλιο για το σχέδιο αυτό του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή σας ε, να παρακολουθεί όσο το δυνατόν πιο στενά την εξέλιξη αυτού του φιλόδοξου και πολύπλοκου σχεδίου, όπως γνωρίζετε, αλλά ταυτόχρονα και πολύ συναρπαστικού. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε πλέον να το χωρίσουμε το ε, πρόγραμμα θα προχωρήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βέβαιο αυτή τη στιγμή. Από την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ, είχαμε μία σειρά από εξελίξεις ε, και νέα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, για την πρωτοβουλία αυτή. Καταρχάς, προχώρησε πάρα πολύ το θέμα του κτηρίου ε, στο οποίο θα στεγάζεται το μουσείο. Όπως γνωρίζετε πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο ε, σχέδιο. Αρχικώς υπήρχε μια γενικότερη ενημέρωση ε, σε όλο τον κόσμο των μουσείων και σε ομάδες αρχιτεκτόνων και είχαμε ως αποτέλεσμα να έχουμε πάνω από 100, 130 περίπου μελέτες, ε, ε, συγγνώμη, μελετητικά γραφεία, τα οποία ήρθαν σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες αφού έλαβαν ε, τις πληροφορίες, περίπου 30 εξεδήλωσαν ένα πιο συγκεκριμένο ενδιαφέρον και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο. Και οι 30 αυτές προτάσεις ε, μελετήθηκαν από ανθρώπους φυσικά που ε, γνωρίζουν τα θέματα αυτά εντός του Κοινοβουλίου και έχουμε 12 πλέον σε επίπεδο προσχεδίου. 12 προτάσεις από όλες τις γωνιές της Ευρώπης και από αυτές τις 12 προτάσεις έγινε μια διαδικασία επιλογής από ιδιαίτερα ικανούς ε, κριτές, κάποιου από τους καλύτερους αρχιτέκτονες της Ευρώπης και καταλήξαμε σε τρεις από τις τρεις ε, στις δύο προτάσεις και από τις δύο στη μία. Φτάσαμε λοιπόν στο πλέον ένα σχέδιο Σες Εμορέλ ονομάζεται το σχέδιο αυτό. Πρόκειται για μια γαλλική ομάδα η οποία ε, όμως ε, ε, συμμετέχει με μια γερμανική και βελγική ομάδα ταυτόχρονα. Αυτό ήταν ε, κοινοπραξίες ε, εν γέννη προτάσεις που είχαμε. Οι κύριοι όμως της πρότασης είναι η γαλλική ομάδα είναι αυτοί που έκαναν και το πετί του Παρισιού και έγιναν και κάποια από τα πιο σημαντικά και πιο ενδιαφέροντα μουσεία από πλευράς τους όπως το Μουσείο της Τουλούζ το κτίριο, όπως γνωρίζετε, είναι το κτίριο Ιστμάν που βρίσκεται εδώ απ' έξω. Εκεί θα στεγαστεί το μουσείο. Είναι ένα κτίριο για το οποίο άκουσα διστάμενες απόψεις. Εμένα μου φαίνεται ένα αρκετά ενδιαφέρον ε, ε, σύγχρονο κτίριο. Σε αυτό το κτίριο λοιπόν, το οποίο έχει μορφή... Ε, σε ένα σχήμα γιου και εκεί στο κενό τέλος πάντων του σχήματος αυτού θα στεγαστεί το μουσείο. Υπάρχει το σχέδιο λοιπόν και βάσει αυτού θα προχωρήσει το μουσείο. Και τέλος υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο, είναι το στοιχείο του προεπολογισμού Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε για το 2012 13 εκατομμύρια ευρώ κονδύλιο, πρόκειται για σεβαστό ποσό φυσικά. Εγκρίναμε τα 11 εκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στον προϋπολογισμό και 2 εκατομμύρια από το αποθεματικό. Και για το 2013 στις ε, προβλέψεις που έχουν εξελίξει δεν έχουν κατατεθεί σχετικές τροπολογίες βέβαια εκτός από κάποιες πολύ μειονοτικές ομάδες ή από μεμονωμένους ευρωβουλευτές για το 2013 λοιπόν προβλέπεται ένας προϋπολογισμός 11 εκατομμυρίων ευρώ και για το 2014 4 εκατομμύρια ευρώ Αυτά λοιπόν προβλέπονται προς το παρόν αν και πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά έχω όλο και περισσότερες ανησυχίες και αμφιβολίες ε, για το κατά πόσον θα ε, υπάρξουν εγγένεια του οίκου της Ευρωπαϊκής Εστερίας το ε, πρώτο εξάμεινο του 2014, δηλαδή πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να σας επισημάνω ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος και ως προς το περιεχόμενο του οίκου της ευρωπαϊκής ιστορίας. Υπάρχει πλέον μία τεχνική ομάδα. Έχουν επιλεγεί οι επικεφαλής του προγράμματος. Η κυρία Φοκνάλη θα είναι η Γενική Διευθύντρια του Μουσείου, η οποία είναι εδώ σήμερα και νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή να έρθει και εδώ στην Επιτροπή σας για να σας εξηγήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να συζητήσει μαζί σας το περιεχόμενο. Ε, πέραν της Γενικής Διευθύντριας, η οποία επελέχθηκε μετά από μια μακρά διαδικασία και περίπλοκη επίσης, Θεωρώ βέβαια ότι ήταν ιδιαίτερα διάφανη διαδικασία, αλλά όπως γίνονται τα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας δηλαδή πάντα υπόψη ότι είχαμε πάμπολους υποψηφίους, έπρεπε να ακούσουμε τους μεν και του δε, αρχικώς ε, χρειάστηκε να γίνει μια πρώτη επιλογή μέσω βιογραφικών σημειωμάτων, κάτι το οποίο αφήνει και κάποια πικρία, διότι απορρίπτονται άτομα τα οποία θα μπορούσαν να μας ε, δώσουν πολύ σημαντικά προσόντα, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν η διαδικασία. Τελικώς καταλήξαμε σε 8-10 άτομα και από εκεί και πέρα έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση στην ε, Επιτροπή Επιλογής ε, και τελικώς καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση. Υπάρχει και μία ομάδα 18 ιστορικών οι οποίοι επίσης ε, προσελήφθησαν. Ε, πρόκειται για άτομα με μεγάλη εμπειρία από 13 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, από όλες τις άκρες της Ευρώπης, από το βορρά, τον νότο και φυσικά ο καθένας με την ε, εξειδίκευση που απαιτείται στη συνέχεια για το μουσείο. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης, το οποίο θα ήθελα να σταθώ, και ορισμένες φορές δεν αναφέρεται από την ομάδα του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ε, είναι το γεγονός ότι εγγενιάστηκε το Παλαμερτάριουμ που είναι το κέντρο των επισκεπτών και θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ε, εμπειρία αρκετά επιτυχημένη και δεδομένου ότι έχουμε και αυτό το αιώραμα για τον οίκο της Ευρωπαϊκής ε, Ιστορίας είναι δεδομένο ότι το σχέδιο του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα πρέπει να λάβει υπόψη το Παρλαμεντάριο και να προσαρμοστεί σε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει και με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο δείχνει πώς ε, είναι δομημένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις ε, και να μην εκτίθενται και στις δύο ε, <clears throat> περιπτώσεις τα ίδια πράγματα αλλά να γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα όπως γνωρίζετε ε, και εσείς έχουμε την ίδια πρόθεση να ενημερώνουμε και να ε, διαβιβάζουμε στους πολίτες μας πώς είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ποια είναι η ευρωπαϊκή ε, ταυτότητα και πώς προχωράει η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάποια στοιχεία του Παρλαμεντάριου. Για παράδειγμα, όλο ο μηχανισμό τη πολυγλασία, ο οποίο είναι εξαιρετικό. Δεν ξέρω ποιοι από εσά έχουν επισκεφθεί το Παρλαμεντάριο. Όσοι δεν το έχετε επισκεφθεί, σα καλώ λοιπόν να πάτε να το δείτε, διότι το θέμα τη πολυγλωσία είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά κομμάτια μπορεί να μπουν τέσσερις πολίτες από τέσσερις διαφορετικές χώρες που μιλούν μια διαφορετική γλώσσα από τις 23 επίσημες γλώσσες που θα γίνουν 24 με τα κροάτικα σύντομα. Ο καθένας λαμβάνει μια συσκευή και μπορούν να προχωρούν μαζί και ο καθένας να ακούει. Άλλο στα γερμανικά, άλλο στα ισπανικά, άλλο στα ελληνικά και άλλο στα ρουμάνικα ή τα σλοβένικα. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας και φυσικά... Ε, όλα όσα θα μάθουμε από την ε, διαδικασία του Παρλαμεντάριου και οποιαδήποτε βελτίωση μπορούσαμε να έχουμε εκεί, ε, σίγουρα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Προς το παρόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα σας ενδιαφέρει ίσως να ακούσετε είναι και το γεγονός ότι αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε δύο πράγματα. Πρώτον, πώς ακριβώς θα έχει το μουσιακό περιεχόμενο του οίκου της ευρωπαϊκής ε, ιστορίας, έχοντας πάντα ως ε, σημαντική πηγή έμπνευσης ε, το House The Deutsche που έχει και αυτό το εξαιρετικό μουσείο της Βόνης αλλά και το μουσείο της Λιψίας το οποίο επισκεφθήκαμε και φυσικά λαμβάνονται υπόψη και κάποιες πρωτοβουλίες που ξεκινούν ε, ε, μέσω αυτής της δραστηριότητας και στο Βερολίνο. Το τι θα περιλαμβάνει λοιπόν το μουσείο είναι κάτι το οποίο εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι τεχνικοί μας, οι εμπειρογνώμονές μας και πρέπει να σας πω ότι αυτοί που είμαστε στη διεύθυνση του όλου προγράμματος από πλευράς Προεδρίου δεν θελήσαμε να παρέμβουμε διότι θεωρούμε αυτής εξ αρχής ότι οι ιστορικοί και εμπειρογνώμονε είναι αυτοί που θα ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Βεβαίως κάποια στιγμή θα πρέπει να παρέμβουμε κι εμείς λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι ε, συμφωνούμε όλοι επί της αρχής. Δηλαδή το να έχουμε ένα μουσείο 4.000 τετραγωνικών μέτρων ε, που θα έχει μία μόνιμη έκθεση και ταυτόχρονα να έχουμε και 8.000 τετραγωνικά μέτρα 800 συγγνώμη, τετραγωνικά, τα οποία θα έχουν ε, περιοδικές εκθέσεις. Ερχόμαστε σε επαφή και με διάφορα κέντρα και ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, μουσεία, ε, πανεπιστήμια, ε, του πολιτισμού, οίκους Ευρώπης, διάφορα δηλαδή ιδρύματα, τα οποία ελπίζουμε ε, να συνεχίσουν να δίνουν το ενδιαφέρον που δείχνουν και θα πρέπει να συσχετιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο με το όλο ε, ε, πρόγραμμα περιοδικές εκθέσεις που γίνονται εδώ και θα μπορούσαν ίσως να, να πάνε και αλλού ή οτιδήποτε μας προτείνουν όλοι αυτοί οι συνομιλητές μας που θα μπορούσαμε να το φέρουμε εδώ λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει και αυτός ο επιπλέον χώρος διαθέσιμος. Ε, έχουμε λοιπόν τα εξή. Καταρχά, διαφυλάξαμε ε, ότι δεν υπάρχουν προσκόμματα ω προ τον προπολογισμό και μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τώρα λοιπόν προσπαθούμε να δούμε πώ θα έχει το ε, επιστημονικό, επιτρέψτε με τον όρο, ή ακαδημαϊκό περιεχόμενο των εκθέσεων και της μόνιμης και των περιοδικών εκθέσεων και επίσης υπάρχει και μια διαδικασία την οποία θα ήθελα να αντιμετωπίσω όσο το δυνατόν πιο διπλωματικά, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι κάποιους εξημών μας εξέπληξε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να λάβουμε τις απαραίτητες άδειες για να γίνουν τα έργα κάποιοι από εμά που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα αυτά ε, είχαμε την εντύπωση ότι όταν υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχουν και αρχιτέκτονες οι οποίοι διψούν να προσφέρουν, ε, η άδεια είναι αυτόματη. Τελικώς όλα αυτά δεν είναι αυτόματα βέβαια. Ε, το βελγικό κράτος έχει μια πολύ περίπλοκη δομή. Βέβαια δεν είναι πιο περίπλοκη από οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή χώρα, να μην σας πω για τη χώρα μου ας πούμε, αλλά σίγουρα είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Δεν έχουμε έναν συνομιλητή απέναντί μα, αλλά έχουμε τέσσερις ή πέντε συνομιλητές. Υπάρχει το βελγικό κράτος, ο συνομιλητής ε, ε της περιφέρειας ή της κοινοτητα αν θέλετε, ε, ο δημο Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν γνώριζε σχεδόν κανείς. Υπάρχει η Επιτροπή ε, Προστατευόμενων Χώρων διατηρητέων κτηρίων φαντάζομαι. Υπάρχουν δηλαδή και διάφορα πρόβλεπτα στοιχεία. Ε, παραδείγματος χάρη το πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του ε, σε κάποια στοιχεία του προγράμματος. Ε, μπορεί να υπάρχει και μία καθυστέρηση δύο μηνών για παράδειγμα για να εγκριθεί κάτι τέτοιο. Όλα αυτά φυσικά δεν μπορούμε να τα ζητήσουμε ταυτόχρονα. Πρέπει να λαμβάνουμε την άδεια για το ένα και σιγά σιγά να προχωρούν τα υπόλοιπα. Όπω προχωρούν τα διάφορα στοιχεία δηλαδή έχουμε το ένα εμπόδιο στο άλλο. Οι βελικές αρχές από την άλλη μεριά πρέπει να πω ότι είναι ενθουσιασμένες με το σχέδιο αυτό. Προφανώς στην καρδιά της πρωτεύουσα της χώρας θα δημιουργηθεί ένα μουσείο ε, εμβέλειας, εμβέλειας, μεγάλης εμβέλειας, αρχιτεκτονικής και μουσιακή εμβέλειας, οπότε είναι προφανές ε, οι βελικές αρχές να είναι υπέρ της δημιουργίας του. Πολύ δε περισσότερο που δεν τους ε, ζητούμε ούτε ένα ευρώ. Βέβαια, από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι ανησυχούν διότι το μουσείο θα, βρε, θα βρίσκεται στο πάρκο Λεοπόλτ το οποίο γενικότερα έχει αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Συνεπώς, τίθενται διάφορα τεχνικά ζητήματα. Δεν μπορούμε να ανέβουμε σε αυτό το ύψος γιατί θα καλύψουμε τη θέα του άλλου κτηρίου που βρίσκεται από πίσω κλπ. κλπ. Είναι θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εμφανιστούν και σε οποιαδήποτε από τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το στάδιο. Το μουσείο θα, θα δέχεται τρεις τύπους επισκεπτών. Πρώτον, Ευρωπαίοι επισκέπτες. Μέσα σε αυτούς τώρα θα έχουμε αυτούς που θα έρχονται από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτούς που θα προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά θα έχουμε και ένα άλλο τύπο επισκεπτών που θα είναι όλες αυτές οι ομάδες που προσκαλούμε εμείς πολλές χιλιάδες κάθε χρόνο και μετά με μονομενοι επισκέπτες, τουρίστες της Βρυξέλλες για παράδειγμα. Και μετά θα υπάρχουν και πολλοί που δεν θα είναι καν Ευρωπαίοι. Γιατί το μουσείο θα πρέπει να απευθύνεται και στους μη Ευρωπαίους. Θα ε, φτάνουν και Αφρικάνοι και Κινέζοι και Ιαπωνέζοι και Λατινοαμερικάνοι που δεν είναι Ευρωπαίοι ούτε καν σκέφτονται να γίνουν Ευρωπαίοι. Αλλά τους ενδιαφέρει και αυτούς η συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό το μουσείο. Ένα θαύμα ε, σε μια Ήπειρο που για πολλούς αιώνες χαρακτηριζόταν από συγκρούσεις. Μια Ήπειρο στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, έχουν ε, βλαθεί περισσότερο από ότι σε οποιαδήποτε άλλη ήπειρο. Και σε, μέσα σε μερικές δεκαετίες, δύο-τρεις δεκαετίες, αυτή η ίδια ήπειρος γίνεται παράδειγμα ολοκλήρωσης και μια βιτρίνα αξιών ε, που τη χάνουν εκτίμηση πολύ περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Από ό,τι οπουδήποτε αλλού. Συνεπώς δεν ενδιαφέρονται μόνο οι ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χώρες όπως η Ρωσία ή η Τουρκία. Μπορώ να σας πω ότι ενδεχομένως εκφράζουν και περισσότερο ενδιαφέρον από ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θεωρούν τον εαυτό τους τμήμα της ευρωπαϊκής ιστορίας και ανησυχούν για το πώς θα εμφανιστεί ο δικός τους ρόλος στην ευρωπαϊκή ιστορία. Θα ληφθεί υπόψη η Ρωσία, η Τουρκία και πώς. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, Πω, τι ρόλο θα παίζει σε αυτό το μουσείο. Ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αναρωτιόνται πώς θα εμφανίζονται και πώς θα παρουσιάζονται στο μουσείο. Οι χώρες επίσης που ήταν απικίες ευρωπαϊκών χωρών. Πιο πολλές επαφές έχω με αυτές τις χώρες παρά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται πιο πολύ σε επαφή μαζί μας. Έχω την εντύπωση ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το project αυτό δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ενθουσιασμό που αντιμετωπίζεται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα βέβαια δεδομένου ότι έχουμε εξασφαλίσει τη συνέχεια του project αυτού, ίσως δεν, έχουμε, δεν το έχουμε δημοσιοποιήσει τόσο πολύ όσο θα χρειαζόταν. Ο κύριος ε, Πέτερινγκ ήταν ο εμπνευστής του σχεδίου αυτού. Ε, είχαμε διοργανώσει μια συνέντευξη τύπου στην οποία εγώ δεν κατάφερα να ε, φτάσω διότι ε, έπεσε μερικούς ορόφους στο ασανσέρ που με μετέφερε. Ε, βρέθηκε ο, κύριος Πέτερινγκ μόνος του λοιπόν, ε, εμείς οι υπόλοιποι μαζί με την κυρία Ζανίκη από την ομάδα σου ε, ήμασταν απομονωμένοι, κλεισμένοι, μπλοκαρισμένοι σε ένα σανσέρ για δυόμιση ώρες. Και αυτό αποτελεί τμήμα της, ιστορίας, της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτά. Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σας είμαι πρόθυμος να την απαντήσω. Θα ήταν ε, ενδιαφέρον μέλη της Επιτροπής σας να παρακολουθούν τακτικά τις εξελίξεις. Ο Πέτερινγκ, εγώ ίδιος και άλλα μέλη του προεδρίου σκοπ Επίμως δεν έχουμε ως τώρα συμμετάσχει στην επιστημονική συζήτηση, στον επιστημονικό διάλογο, ε, του οποίου επικεφαλής είναι η μελλοντική διευθύντρια του μουσείου. Πλην όμως κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς να συμμετάσχουμε ως κοινοβούλιο. Γιατί, γιατί η ευθύνη τελικά δεν θα είναι ευθύνη της επιστημονικής ομάδας, θα είναι μια πολιτική ευθύνη του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, συναδέλφων, ενδεχομένως ας πούμε αυτής της Επιτροπής ή οποιασδήποτε άλλης Επιτροπής θα ασχοληθεί ε, με το μουσιακό περιεχόμενο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Άγχελ. Έχουμε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο και ιδιαίτερα πολιτιστικό σχέδιο που έχει πολλά να κάνει με την καθημερινή μας ζωή στην Ευρώπη και μας ενδιαφέρει όλους. Λοιπόν, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο της Ευρώπης, της ιστορίας της Ευρώπης και γι' αυτό και ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν πρέπει λοιπόν να παραμελήσουμε τίποτα από την ιστορία μας αυτή και αντίθετα από ό,τι πιστεύουν πολλοί δεν είναι ένας ανταγωνιστής του Παρλαμεντάριου, είναι ένα διαφορετικό εγχείρημα, πρόκειται για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό από το, πλαν, που έχει να κάνει με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα μεγάλο πολιτιστικό σχέδιο και πιστεύω ότι εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να το υποστηρίξουμε πλήρως, το έχουμε πράξει πλήρως μέχρι στιγμής. Η κυρία Παλιαδέλη εξάλλου έρχεται και από τον τομέα των μουσείων και της προστασίας μνημείων την ενδιαφέρει διατήρηση πολιτιστική κληρονομιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα πολύ καλό δρόμο για τα θέματα αυτά και δεν θέλουμε να κάνουμε ένα σχέδιο σε μικρή κλίμακα, αλλά έχουμε εμπλέξει εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη και έχει γίνει μια επιλογή διάφανη όλων αυτών των εμπειρογνωμών. Δεν είναι ένα γαλλικό ή γερμανικό εγχείρημα, είναι κάτι το οποίο καλύπτει όλη την Ευρώπη. Ήδη άτομα από την Πολωνία, παραδείγματος χάρη, ήρθαν και συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο ο Πολωνός Αντιπρόεδρος επιπλέον, μάλλον υπάρχει ένας Πολωνός στο Προεδρείο της ε, ομάδας αυτής που επεξεργάζεται το σχέδιο. Όλα αυτά επίσης και οι υπεύθυνοι για τα καλλιτεχνικά θέματα που θα πρέπει να δούνε τι ακριβώς θα εκτίθεται σε αυτό το κτίριο του οίκου της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Εν πάση χρειάζεται να υποστηρίξουμε όλους αυτούς που έχουν το δύσκολο αυτό έργο επιλογής. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ για το έργο σας. Θα πρέπει να είμαστε πάντα στο προσκήνιο και την πρωτοπορία δεν χρειάζεται να εξηγήσω στους συναδέλφους μου γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το εγχείρημα του οίκου της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να μιλάμε μονάχα για την οικονομική κρίση και τη χρηματοδότηση του πολιτιστικού τομέα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την πολιτιστική κληρονομία ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής ιστορίας και μπορούμε χωρίς καμία ανησυχία να τονίσουμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Έχω γνωρίσει και εγώ ίδια πόσο δύσκολο είναι να επιτύχει κανείς κάτι τέτοιο όταν είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα, όταν είναι τόσο δύσκολο το να κάνει κανείς τις σωστές επιλογές. Είναι σημαντικό λοιπόν που έχει ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα και ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω καθυστέρησεις και θα υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα πω. Κύριε Μιγκάλσκι, έχετε το λόγο. E, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Μιγκάλσκι. Κάποια σχόλια θα ήθελα να κάνω και να θέσω και ορισμένα ερωτήματα προς τον κύριο Μαρτίνεθ. Το πρώτο μου σχόλιο αφορά το γεγονός ότι στο τέλος της παρουσίασής σας, κύριε Μαρτίνεθ, είπατε κάτι το οποίο ίσως δεν θέλατε να το πείτε. Είπατε ότι αυτό θα είναι ένα μουσείο που θα δείχνει το θαύμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πώς δηλαδή η Ευρώπη έχει καταφέρει να ενοποιηθεί στις τελευταίες δεκαετίες και τώρα αυτό έχει γίνει πραγματικότητα. Εγώ τώρα δεν καταλαβαίνω αν πρόκειται για οίκο ευρωπαϊκής ιστορίας ή για ένα οίκο ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι σαφές για μένα. Ένας γνωστός Άγγλος φιλόσοφος ο Μπέρχαρτ είπε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούμε Όκα μάλλον είπε ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε περαιτέρω ε, οντότητες από ό,τι είναι απαραίτητο. Η Ευρώπη έχει μια ιστορία που ανατρέχει σε χιλιάδες ετών, σε χίλια χρόνια τουλάχιστον. Πώς μπορούμε να συμπυκνώσουμε όλη αυτή την ιστορία σε 800 μονάχα ψωροτετραγωνικά μέτρα. Πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για επιλογή. Και αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι πολιτικές και όχι καλλιτεχνικές αποφάσεις. Όσο μεγάλο και να είναι αυτό το μουσείο λοιπόν θα πρέπει να περιοριστούμε από τις διαστάσεις του. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ένα είδος εγκλήματος αδικοπραξίας κατά της ευρωπαϊκής ιστορίας. Κατανοώ ότι ένα μουσείο για την ιστορία της Γερμανίας ή της Πολωνίας ή της Ισπανίας θα ήταν κάτι πιο απλό. Θα μπορούσε σε ένα κτίριο να συμπεριληφθεί, αλλά εμεί δεν μπορούμε σε ένα κτίριο να συμπεριλάβουμε στοιχεία της ιστορίας όλης της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Γι' αυτό έχω κάποιες αμφιβολίες. Και τώρα τα συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον κύριο Ματίνες. Πόσο θα κοστίσει η συνολική δημιουργία αυτού του μουσείου. Είπατε πόσα εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται στον προπολογισμό. Αλλά ποιο είναι το συνολικό κόστος της δημιουργία αυτού του μουσείου, θα ήθελα να ξέρω. Δεύτερο ερώτημα. Είπατε ότι υπάρχουν 18 ιστορικοί οι οποίοι επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή το σχέδιο αυτό από 13 χώρες. Δηλαδή άλλα 14 κάτι μέλη δεν εκπροσωπούνται σε αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή από του ιστορικού. Κάποιε χώρε μπορεί να εκπροσωπούνται από περισσότερο από περισσότερους του ενός ιστορικούς. Άλλες χώρες δόλος. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος είναι ο κατάλογος των ιστορικών για να δούμε ποιοι είναι. Ευχαριστώ κύριε Μιγκάσκι. Είναι όλα απόλυτα διάφανα. Υπάρχει και ένας ε, Πολωνός ιστορικός αλλά δεν νομίζω ότι δεν είναι σε θέση να κατανοήσει το σύνολο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτό ισχύει για όλους και για τους Πολωνούς και τους Γερμανούς. Δεν χρειάζεται ένας Πολωνός ιστορικός για την πολωνική ιστορία. Αυτό θα ήταν κάπως μικρόπνο. Η κυρία Κάλεμπαχ. Κάλεμβερτ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ πιστεύω ότι οι ιστορικοί δεν, είναι τόσο, δεν έχουν τόσο περιορισμένους ορίζοντες ώστε να μην μπορούν να κοιτάξουν πέρα από τα εθνικά τους στοιχεία. Νομίζω ότι είναι λογικό να πιστεύουμε ότι η ομάδα αυτή ιστορικών έχει αρκετά ανοιχτού ορίζοντες και θέλουν να βρουν τον πιο λογικό τρόπο να παρουσιάσουν τα στοιχεία αυτά της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι γεγονός βέβαια ότι έχουμε περιορισμένο χώρο 4.000 τετραγωνικά μέτρα και άλλα 800 για προσωρινές εκθέσεις αυτό το θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε διάφορες εκθέσεις που δίνουν μια ιδιαίτερη έμφαση και προβολή σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζω απόλυτα αυτή την πρόταση που έχει γίνει ώστε κάποια στιγμή σε μια πεταγενέστερη ευκαιρία να ακούσουμε και τη, αυτά που έχει να μας πει η διευθύντρια αυτού του μουσείου για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς θα μπορέσει να παρουσιαστεί η, η πολύπλευρη φυσικά ευρωπαϊκή ιστορία σε 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Δεν θέλουμε να περικόψουμε τίποτα, αλλά φυσικά δεν μπορούμε όλα να τα παρουσιάσουμε μόνο με 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Και ίσως θα μπορούσε ο κύριος Μαρτίνε να μας παρουσιάσει πιο λεπτομεριακά τα θέματα αυτά, ίσως σε μια μικρή ομάδα από την Επιτροπή μας. Γιατί εμείς έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ για το τι θα σήμαινε 20 της ευρωπαϊκής ιστορία και με τον κύριο Ήβαρ είχαμε συνεργαστεί για μια θεματική προσέγγιση για τα θέματα αυτά για να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε κάπως την προσέγγιση αυτή χωρίς να πούμε εντάξει τα κόβουμε αυθαίρετα και ξεκινάμε το 1970 και μόνο από εκεί και πέρα λειτουργούμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παιδαγωγική πτυχή ενός τέτοιου μουσείου και θα ήταν χρήσιμο να σκεφτούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά και ο επισκέπτης. Επίσης για τα οικονομικά θέματα, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο μα ενδιαφέρει. Ξέρω ότι έχουν γίνει συζητήσεις για το κόστος λειτουργίας του μουσείου στο μέλλον. Έχουμε από τη μια μεριά το κόστος δημιουργία το οικονομικό και διαρθμιστικό κόστος, αλλά η άλλη πλευρά του νομίσματο είναι πόσο θα είναι το κόστος λειτουργίας, το λειτουργικό κόστος του μουσείου στη, στο μέλλον και εδώ υπάρχει και μια συζήτηση για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμμετάσχει στην κάλυψη του λειτουργικού κόστους γιατί η ευρωπαϊκή ιστορία προφανώ δεν είναι μονάχα κάτι που εμπλέκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί είμαστε ένα σημαντικό κομμάτι τη ευρωπαϊκή ιστορία. Θα ήταν χρήσιμο όμω να μην προέρχονται τα κονδύλια μόνο από τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά να συμμετέχουν αναλογικά και τα άλλα θεσμικά όργανα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πρόοδο να μας ε, περιγράψετε για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέγει η πρόοδος. Εμείς δίνουμε τα λεφτά. Οι, τα άλλα θεσμικά όργανα μέχρι στιγμής δεν έχουν συμβάλει, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και αυτή τη δυνατότητα. Μπορούμε, να το κάνουμε και εθελοντικά, εάν το θέλουμε. Κύριος Τέκες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Αντιπρόεδρε. Και εγώ, ως Αντιπρόεδρος είχα λάβει μέρος σε συνεδριάσεις του Προεδρείου όπου ο κύριος ε, Πέτερινγκ μας είχε περιγράψει εν λεπτομερία όλα τα στοιχεία αυτού του εγχειρήματο του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα πράγματα τώρα προχωρούν εμείς τώρα ως Επιτροπή Πολιτισμού είναι τμήμα και του δικού μας εγχειρήματος να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Γιατί μας ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή ενότητα και ολοκλήρωση. Όταν βρισκόμαστε σε μία φάση οικονομικής κρίσης δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και τον ρόλο που παίζει η κουλτούρα στην καθημερινή μας ζωή. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ και θέλω να εκφράσω και την ευαρέσκειά μου προς τον κύριο Μαρτίνες για όλα αυτά τα οποία μας έχει αναφέρει. Και ίσως θα έπρεπε ορισμένοι τομείς οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί μέχρι τώρα να έρθουν στο προσκήνιο και η Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να συμβάλλει και να εξασφαλίσει ότι θα γίνει η σωστή επιλογή. Έχουμε το θέμα των ολοκληρωτικό καθεστώτος στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ο κύριος Μαρτίνες και αυτός έρχεται από μια χώρα όπου για ένα χρονικό διάστημα υπήρξε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Και εγώ είχα μια αντίστοιχη εμπειρία και υπήρξαν ολοκληρωτικές δικτατορίες και στην Ανατολική αλλά και στη Δυτική Ευρώπη. Και φυσικά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το φαινόμενο της δικτατορίας στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με τις δικτατορίες στη Δυτική ή στην Ευρωπαϊκή ε, Ευρώπη. Κάθε δικτατορία είναι δικτατορία. Και τώρα έχουμε ξεπεράσει βέβαια αυτή τη φάση ολοκληρωτικών καθεστώτων, αλλά δεν πρέπει να λησμονήσουμε αυτά τα στοιχεία. Σε σχέση τώρα με το κτίριο, έχουμε δημιουργήσει στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλλον την πλατφόρμα αυτή για την ιστορική μνήμη. Και η κυρία Γκάλ είχε αντιμετωπίσει το θέμα αυτό στο παρελθόν. Θα ήθελα και αυτό να ληφθεί υπόψη. Ψήφισαμε ήδη την έκθεσή μου σε σχέση με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και εκεί στα αγγλικά λέει το κείμενο ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε οποιαδήποτε ιστορική μελέτη τα πρώην, ε, τα πρώην ολοκληρωτικά καθεστώτα της ε, Ευρώπης ως πηγή διδαγμάτων. Πρέπει να λάβουμε επίσης και την χριστιανική διάσταση της Ευρώπης. Ζούμε σε, μια, σε ένα κοσμικό κράτος. Τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα τους είχαν περάσει σε μια διάσταση αθεϊστικής κοινωνικής ζωής. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχει και η θρησκευτική συνείδηση σαν στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ένα τρίτο σημείο το οποίο πολλές φορές τη χάνει, το παραγνωρίζει κανείς, είναι η σύνολη προβληματική των μειωνοτικών ομάδων. Σχεδόν κάθε έβδομος Ευρωπαίος πολίτης ανήκει σε μία μειονότητα. Οι μειονότητες λοιπόν είναι σημαντικές και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό για μας ως Ευρωπαίους. Λέει ο κ. Μιγκάλσκι ότι στην ομάδα των ιστορικών δεν εκπροσωπούνται <clears throat> όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχει ο κίνδυνος να, κρίνει, να κριθεί κάθε κράτος μέλος από πολλά κράτη-μέλη να κρυθούν από ανθρώπους που δεν προέρχονται από τις χώρες αυτές. Μα δεν μπορούμε να ξέρουμε όλα. Κανείς δεν ξέρει και την τελευταία λεπτομέρεια του τι έχει συμβεί στην τελευταία περιφέρεια και γωνιά της Ευρώπης αυτά τα οποία έγιναν παραγωγικά στην Τρανσιλβανία, στη Ρουμανία. Από τον 6ο ε, αιώνα ήδη υπήρχε μια ιδιαίτερη κατάσταση, υπήρχε το 16ο αιώνα, συγγνώμη, υπήρχε ήδη μια ρύθμιση που εξασφάλιζε την ανεξιθρησκεία, το γεγονός ότι όλες οι ομολογίες και τα δόγματα της χριστιανικής εκκλησίας μπορούσαν να συνεπάρχουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα επίσης σε σχέση με την έννοια της κεντρικής Ευρώπης. Τι είναι η κεντρική Ευρώπη. Πού αρχίζει, πού σταματάει η κεντρική Ευρώπη, ποια είναι η διάσταση τη κεντρική Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα νομίζω ότι πρέπει να τα λάβει υπόψη και η Επιστημονική Επιτροπή. Προφανώ όλα αυτά θα, κάποιο, παίζαν κάποιο ρόλο. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε του εμπειρογνώμονε να συζητήσουμε με τα θέματα αυτά. Βέβαια, κανείς δεν θα είναι ποτέ απόλυτα ικανοποιημένος. Αλλά κύριε Τόκε, είμαι σίγουρος ότι οι επιστημόνες που βρίσκονται σε αυτή την Επιτροπή σίγουρα θα χρησιμοποιήσουν τις ε, γνώσεις τους όχι για να παρουσιάσουν μόνο μια γερμανική ή μια γαλλική οπτική γωνία, αλλά για να δουν τι έχει γίνει και πώς έχουν εξελιχθεί τα θέματα αυτά σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα, όλες αυτά τα θαυμάσια ζωγραφισμένα μοναστήρια στη Ρουμανία, στο Ζήμπιο και σε άλλα μέρη. Πιστεύω λοιπόν ότι οι ιστορικοί θα μπορέσουν να εκτιμήσουν όλα αυτά τα στοιχεία και αυτή είναι μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει νόημα να την κάνουμε με του εμπειρογνώμενους. Είναι θαυμάσιο συνάδελφο και θαυμάσιος άνθρωπο ο κ. Μαρτίνες, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν είναι το δικό του καθήκον να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα αυτά, δεν μπορεί να ξέρει όλε αυτέ τι λεπτομέρειε. Αυτά είναι η υπευθυνότητα μονάχα μια ομάδας επιλεγμένων ιστορικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά και ίσω θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια επαφή μαζί του. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και για αυτά τα οποία είπατε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας επισημαίνετε γιατί βρίσκονται πολύ κοντά στην καρδιά μας όλα αυτά. Κυρία Βεργία, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ για την τακτική ενημέρωση που μας παρέχει για αυτό το τόσο όμορφο και ενδιαφέρον σχέδιο. Νομίζω ότι αν δούμε την Ευρώπη από το πρίσμα της ιστορίας μας επιτρέπει, θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα όπως οι εθνικισμοί για παράδειγμα. Ε, διότι με αυτόν τον τρόπο σχετικοποιούμε τα πράγματα. Η ιστορική οπτική γωνία βάζει πολλά πράγματα στη θέση τους. Ε, διάβασα ένα μικρό βιβλίο τελευταία που δημοσιεύτηκε στη Γαλλία ε, που λέγεται «Οι πρόγονοί μας, οι γαλάτες και άλλες φαντασιώσεις». Ε, νομίζω ότι είναι μια συμπίκνωση όλων αυτών που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο μουσείο. Ασφαλώς και ο κ. Μαρτίνες δεν πρόκειται να απαντήσει όλα τα ερωτήματά μας. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την μελλοντική διευθύντρια του μουσείου. Θα ήθελα να δω ποια είναι η προσέγγιση του γιατί ελπίζω ότι θα μας επιτρέψει να βάλουμε πολλά πράγματα στη θέση τους, ιδιαίτερα και για την θρησκευτική διάσταση, γιατί στο όνομα της θρησκείας στην Ευρώπη ε, έχουμε κατασφάξει, έχουμε κατασφαγή πρώτον μεταξύ μας εμείς οι χριστιανοί και οι χριστιανοί με τους ε, Εβραίους. Οι σφαγές των Εβραίων δεν ξεκίνησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Γαλλία έχουμε ιδιαίτερα φορτισμένη, βεβαρημένη ιστορία σε σχέση με αυτό το θέμα. Ένα ερώτημα έχω. Ε, πολύ συχνά εκνευρίζομαι όταν μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξ ονόματος όλης της Ευρώπης. Συνεπώς, έχω αυτή την αγωνία. Ο κ. Μαρτίνε μα λέει ότι είναι ένα project του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απ' την άλλη μεριά έχουμε πολλέ χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση που έρχονται σε επαφή μαζί μα. Συνεπώ, τι γίνεται η άλλη Ευρώπη, η Ευρώπη που δεν βρίσκεται στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχει τη θέση τη και αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σκούρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μαρτίνες γιατί είναι πάντα συγκεκριμένος και απτός σε αυτά τα οποία μας λέει. Για μένα η ιδέα αυτή του οίκου της ευρωπαϊκής ιστορίας πάντα μου άρεσε ιδιαίτερα. Μας βοηθά μάλιστα να καταλάβουμε και λίγο καλύτερα ποιοι ήμασταν και ίσως και ποιοι θα γίνουμε. Θεωρώ δε ότι κάποια πράγματα λύνονται από μόνα τους. Να σας πω τι εννοώ. Ε, είναι δύνατο να μην διαπιστώσουμε ότι υπήρχε ένα γέννηση μπαρόκ, ε, ε, ρομαντισμός, κοινό ευρωπαϊκός, το οποίο φυσικά από εκεί και πέρα έλαβε την ταυτότητά του, κάποιες συγκεκριμένες επισημάνσεις για κάθε χώρα, αλλά αυτή ήταν η ευρωπαϊκή ιστορία. Ε, ο 19ος αιώνας ήταν, ε, συγγνώμη, 20ος αιώνας ήταν ένας ευρωπαϊκός 20ος ε, αιώνας. Ε, είχαμε δύο παγκοσμίους πολέμους οι οποίοι φυσικά από εκεί και πέρα δημιούργησαν και άλλα δράματα εκτός Ευρώπης. Θα είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και με την Διευθύντρια αλλά και με τους ιστορικούς για να κατανοήσουμε καλύτερα κάποιες πτυχές αλλά τα πανεπιστήμια μας και οι βιβλιοθήκες μας είναι γεμάτα από κείμενα, από βιβλία ευρωπαϊκής ιστορίας, τα οποία ε, περιγράφουν από διάφορες οπτικές ε, των ιστορικών πότε μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή ιστορία. Επομένως υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, ήδη για να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε και κάποιες από τις κριτικές που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να πιέσουμε ιδιαίτερα επί του θέματος αυτού και έχει δίκιο η κυρία Πακ που υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή μας ε, θα πρέπει να είναι ε, αυτή που δίνει το συνεχή αγώνα διότι ο στόχος που έχουμε θέσει είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος και μπορεί να βοηθήσει και εμάς ε, πέρα από τις συζητήσεις που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε, ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε και ποιοι θα είμαστε. Ο κύριο Τάκουλα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, δύο λόγια, πολύ σύντομα και από πλευράς μου, αλλά ίσως και από πλευράς ομάδος μου. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι θα δημιουργηθεί ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας, διότι πρέπει να πούμε ότι ακόμα και οι τελευταίες ευρωπαϊκές δεκαετίες ήταν ε, επιτυχής. Αν δούμε τα θέματα της ολοκλήρωσης, ε, κατανοώ βέβαια ότι υπάρχουν πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν και ίσως δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι πολύ ευνοϊκοί υπέρ αυτού του προγράμματος, αλλά επίσης θα πρέπει να κατανοήσουν πολύ ότι Εάν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση, σίγουρα θα ήταν χειρότερη ε, για την ταυτότητα της Ευρώπης. Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο, σίγουρα θα πρέπει να εμπιστευτούμε τους εμπειρογνώμονές μας. Δηλαδή, αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πώς και με ποιο τρόπο θα πρέπει να δομηθούν ε, οι εκθέσεις και τι αντικείμενα θα πρέπει να περιλαμβάνουν. Ε, κατανοώ ότι υπάρχει φόβος μεταξύ ημών των πολιτικών ε, για το κατά πόσον μπορεί να ε, υπερτονιστούν ε, κάποιες πολιτικές γραμμές ή ιδεολογίες. Αυτό όμως γίνεται γιατί πολλές φορές εμείς πολιτικοί τίνουμε να επιλέγουμε τις απόψεις μας και να τις υπερτονίζουμε. Όταν, για παράδειγμα, ο κύριος Τέκης ε, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντική, ε, σημαντικός ο χριστιανισμός, ε, δεν νομίζω να υπάρχουν πυρογνώμονε και ιστορικοί στην Ευρώπη που θα αποκλείσουν τον χριστιανισμό. Μόνο κάποιοι πολιτικοί για κάποιους λόγους δεν θα θέλανε να αναγνωρίζεται η ιστορία μας και η πολιτιστική μας κληρονομιά ως και τμήμα του χριστιανισμού. Ε, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο χριστιανισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι ιστορικοί βεβαίως δεν θα κάνουν ποτέ κάτι τέτοιο διότι γνωρίζουν την ευρωπαϊκή ιστορία και γνωρίζουν ότι όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και όλη η ευρωπαϊκή εξέλιξη ε, βασίζονται στο χριστιανισμό. πώς οι ουδαϊστικές, ε, χριστιανικές και ελληνιστικές αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εξέλιξης. Θα πρέπει να πω λοιπόν ότι είναι καλό το ε, σχέδιο και φυσικά θα πρέπει να αφήσουμε τις λεπτομέρειες στους ιστορικούς γιατί αυτοί γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και εμείς ως πολιτικοί δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε και να συζητάμε το περιεχόμενο. Υπάρχουν άνθρωποι εγνωσμένου κύρους οι οποίοι ε, σίγουρα θα ασχοληθούν με τα θέματα αυτά με αντικειμενικό και ευρύ τρόπο. και γνωρίζουμε ότι παρά τα σφάλματα και τα κενά που υπάρχουν στην Ευρώπη, η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μια επιτυχής ιστορία. Θα σταματήσω εδώ. Γνωρίζω ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό για κάποιους φίλους μου και χαίρομαι που είναι ιστορικοί αυτοί η μορφώσουν το περιεχόμενο του οίκου της ευρωπαϊκής ιστορίας. Μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε την αντικειμενικότητα. Ο κύριος Κέλλη. Ε, thank uh, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαρτίνεφ για το πολυθετικό του έργο σε ένα ειδικευμένο τρόπο, ε, χώρο που ίσως δεν είναι οικείο σε όλους. Πιστεύω όμως ότι αν, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, μπορέσουμε να εστιάσουμε σε ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και όχι στενές ευρωπαϊκές προσεγγίσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και παρά το γεγονός ότι η ιστορία μας πρέπει να είναι βασισμένη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ιστορία της Ευρώπης μετά από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία λοιπόν 40-50 χρόνια το τι έγινε σε χώρες της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Θέλω και εγώ να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κ. για την σημασία της, ε, του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Εγώ βλέπω να υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παραγνωρίζουν τη σημασία της ε, θρησκείας και επίσης για αυτά που είπε ο κύριος Στάκουλα. Ναι βεβαίως θα πρέπει να αφήσουμε τις λεπτομέρειες τους ε, εμπειρογνώμων, αλλά θα πρέπει να θέσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν και είναι απαραίτητο να έχουμε και εμπιστοσύνη σε αυτό το πλαίσιο. Τελευταία μου παρατήρηση. Εγώ είδα κάποια αρνητικά άρθρα ιδίως σε βρετανικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας για τις ομάδες επισκεπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω εδώ να κάνω δύο παρατήρησεις. Μία, όταν έρχονται οι ομάδες των επισκεπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν προτεραιότητα πρόσβαση στο μουσείο ή όχι. Και δεύτερον πάλι μια σκέψη. Μήπως θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να εάν υπάρχει μια επιδότηση ομάδας των επισκεπτών να είναι υποχρεωτικό να περάσουν λίγο χρόνο στην, ε, στον οίκο της Ευρώπης. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν να ξεπεράσουν μερικές από τις απόλυτα στρεβλωτικές απόψεις που διατυπώνται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες έχουν σαν στόχο να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο σκεπτικισμό, ενώ η επίσκεψη στο μουσείο αυτό θα μπορούσε να τους δώσει μια πιο θετική εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόρης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτίνε εκ βάθους καρδίας. Κατανοώ ότι το πιο δύσκολο πάντα είναι το να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά εμπόδια. Το πιο σημαντικό όμως είναι να καταλάβουμε όλοι ότι είναι μια πολύ θετική ιδέα, κάτι το πολύ φιλόδοξο Κανείς δεν έχει αναλάβει ποτέ το εγχείρημα του παρουσιάσει την ιστορία όλης της Ευρώπης σε ένα μονάχα χώρο. Όσο πιο νωρίς λοιπόν αποφασίσουμε ποιες είναι οι γενικές κατευθύνσεις για το περιεχόμενο των εκθέσεων, τόσο το καλύτερο. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο οδηγεί σε συγκινησιακές προσεγγίσεις. Σίγουρα πρέπει να παρουσιάσουμε την εικόνα και την ιστορία όλη τη Υπήρου, όχι μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ιστορικό γεγονό, αλλά η ιστορία τη Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχαία Ελλάδα, αρχαία Ρώμη, φιλόσοφοι, χριστιανισμό επίπτωση του χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού στην ανάπτυξη του πολιτισμού της Ευρώπης. Βασιλιάδες, αυτοκράτορες, αυτοκρατορίες. Πόσο λοιπόν στενή ή πόσο ευρεία πρέπει να είναι η παρουσίαση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε με τις δικές μας ιδέες. Όσο πιο γρήγορα γνωρίζουμε ποιο είναι το περιεχόμενο του μουσείου, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρος ΠΑΚ. Θα ήθελα η κυρία Φων Φαγκάλ είναι η διευθύνεια του μουσείου βρίσκεται εδώ στο βάθος ε, από την Σλοβενία έρχεται αλλά έχει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων. Έχει λοιπόν επιλεγεί από μια αρμόδια επιτροπή και η Κωνστάς Ευεντζέντς είναι αυτή η οποία εργάζεται για το θέμα αυτό από την επιτροπή μας. Αγαπητέ λοιπόν Άγχελ Ματίνες, έχεις πολλά πράγματα να πεις αλλά παρακαλώ εν συντομία. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω τις απαντήσεις μου σε λίγα σημεία. Καταρχήν κύριε Μιγκάλσκι. Θα ήταν σχετικά εύκολο να φτιάξουμε ένα μουσείο με 27 αίθουσε. Σε κάθε αίθουσα να βάλουμε την ιστορία μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν ακόμα πιο εύκολο αν ζητούσαμε από την κάθε κυβέρνηση να βάλει στην αντίστοιχη αίθουσα την ιστορία της χώρας της. Η πρόκληση είναι να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και έχει δίκιο ο Μιγκάλσκι σε αυτό που λέει. Ε, που ρωτάει αν πρόκειται για την ιστορία της Ευρώπης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την ιστορία της Ευρώπης αλλά κυρίως για την ιστορία της οικοδόμησης της Ενωμένης Ευρώπης. Και αυτή είναι η πρόκληση. Να φτιάξουμε ένα μουσείο για την διαδικασία αυτού του παγκοσμίου θαύματος. Είναι μια έκφραση που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον. Μια διαδικασία στην οποία συμμετείχαν οι άνθρωποι κυρίως. Όχι τόσο οι χώρες, γιατί οι χώρες έχουν εξαφανιστεί, έχουν εμφανιστεί, έχουν μικρύνει, έχουν μεγαλώσει κλπ. Γιατί χώρες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ε, σήμερα δεν υπήρχαν πριν από 100 ή πριν από 70 χρόνια ή πριν από 150 χρόνια. Λίγες είναι οι χώρες οι οποίες υπήρχαν πριν από 150 χρόνια με τα ίδια σύνορα με τα σημερινά. Ίσως τρεις-τέσσερις. Οπότε, Το μουσείο αυτό δεν θα πρέπει να επαναλάβει, ε, να αντιγράψει αυτά που υπάρχουν σε εκατοντάδες άλλα μουσεία. Δηλαδή να λέει Ευρώπη είναι μια ήπειρος που έχει τα εξή ποτάμια, τις εξή θάλασσες και τα εξή σύνορα. Όχι. Θα είναι ένα μουσείο που θα πρέπει να δείχνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Θα δείχνει ότι με βάση συγκεκριμένε αρχές, με βάση συγκεκριμένε αρχές, με βάση τις πολιτικής δραστηριότητας και της ευθύνης που ανέλαβαν οι πολιτικοί σε μια στιγμή μάλιστα που η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα ε, δέχονται έτσι μια πολύ αρνητική συμπεριφορά και ε, ε, έχουν ευτελιστεί στην κοινή γνώμη. Λοιπόν, με βάση τις αρχές της, ε, τη δραστηριότητα και τους πολιτικούς μια Ήπειρος η οποία γνώρισε για εκατοντάδες χρόνια χιλιάδες πολέμους έγινε, κατέστη σύμβολο ειρήνης, σταθερότητας, κοινωνικής προόδρου και ολοκλήρωσης. Και αυτό όλο περιγράφεται με μια λέξη, με δύο λέξεις δηλαδή, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης. Και ό,τι είναι εκτός της ε, και ε, για τις χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί φάρο. Αυτό το βλέπουμε όταν ταξιδεύουμε στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοντέλο για αυτούς για το πώς μπορεί να αντικαταστήσει κανείς ε, τον πόλεμο με την ειρήνη, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σκοτάδι με το φως, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τον ολοκληρωτισμό με τη δημοκρατία. Έτσι είναι η κατάσταση. Τώρα λέτε 4.000 τραγωνικά μέτρα. Ε, εντάξει, ασφαλώς. Ε, εν να σας πω ότι ο επικεφαλής της Ακαδημαϊκής ομάδα είναι ο καθηγητής Μποροτζέη. Ε, νομίζω ότι είναι ένας αξιοσέβαστος ε, Πολωνός, ε, πολύ αποτελεσματικός και πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Ε, καλός φίλος, αλλά πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Οι χώρες έχουν αλλάξει. Εγώ δεν πιστεύω σε κάποια θρησκεία, αλλά έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο II. Και μιλούσαμε για την Πολωνία μαζί του κλπ. Και, και μου είπε κάποια στιγμή Γιατί εγώ του μίλησα για το, τον Μίσκεβιτς, τον μεγαλύτερο Πολωνό ποιητή και μου είπε ο, ο, Πάπας ήταν, γεννήθηκε στη Λιθουανία. Λιθουανός ήταν ο άνθρωπος καταρχήν. Δηλαδή στο Βατικανό το έμαθα ότι ο Μίσκεβιτς είχε γεννηθεί στη Λιθουανία. Τελικά τι είναι ο Μίσκεβιτς, είναι τμήμα της Λιθουανικής ιστορίας ή της Πολωνικής ιστορίας. Όχι, είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Για να μιλήσουμε για τους Ούγγρους. και οι ιστορικοί είναι ίσως οι μόνοι που είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι η ιστορία δεν έχει σύνορα, δεν αναγνωρίζει σύνορα, γιατί τα σύνορα είναι ρευστά. Τώρα, θέσετε και δύο πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις για το κόστος. Περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ το αναφέρει αυτός και ο προπολογισμό. Εντεκάμιση εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος. Μετά, κάποιος μίλησε για το ρόλο της Κομισιόν... ...η οποία έχει αναλάβει τη δέσμευση να συμμετάσχει και πιστεύω θα πρέπει να βρούμε και άλλους χρηματοδότες. Ενδεχομένως το Συμβούλιο ή κάποια Ενδεχομένως ακόμα και ιδιωτικές πηγές που θα ήθελαν να υποστηρίξουν το σχέδιο. Από την άλλη μεριά δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις πριν να ανοίξουμε το μουσείο. Εμείς πρέπει να το ανοίξουμε και άπαξ και το ανοίξουμε ε, θα έρθουν και άλλοι να βάλουν λεφτά δύσκολα κάποιος ιδιώτης θα επενδύσει σε ένα project το οποίο θα εξαρτάται από, την, ε, από τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου. Θα θέλουν να επιβάλλουν τις δικές τους ιδέες. Εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, αλλά ούτε και αυτοί μπορούν να δεχτούν ότι το Κοινοβούλιο μπορεί αύριο να αποφασίσει την ακύρωση του project, ας πούμε. Μετά λέτε 18 ιστορικοί. Προφανώς δεν πρόκειται για ένα ιστορικό ανά μέλος. Και δεν είναι μόνο ιστορικοί, είναι και μουσιολόγοι. Κανένας από αυτούς δεν επελέγει εξαιτίας της ε, εθνικότητάς του. Ε, ούτε ο Πολωνός, ούτε ο Ούγγρος, ούτε ο Γάλλος, ούτε ο Ισπανός επελέγησαν με τέτοιο είδους κριτήριο. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ένα όραμα. Κάποιοι γνωρίζουν βέβαια καλύτερα την ασιατική ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ειδικοί στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι περισσότεροι είναι ειδικευμένοι στον 20ο και 21ο αιώνα, αλλά έχουμε ειδικού και στο μεσαίωνα. Πάνω στο κριτήριο της επικότητας ήταν αυτό που λιγότερο ελήφθη υπόψη. Γνωρίζω κάποιους από αυτούς και ε, χρειάστηκε να, χρειάζεται κάθε φορά να δω την, από πού προέρχονται, γιατί πολύ συχνά θα βρείτε ένα Ισπανό να μιλάει για τις μειονότητες, ένα Ούγγρο να μιλάει για τους θρησκευτικού πολέμους κλπ. Έτσι λειτουργεί η Επιτροπή αυτή. Τώρα, Κυρία Κάλβερτ, ε, πολύ ευχαρίστω, ε, βέβαια, ε, μάλλον θα είναι πολύ χρήσιμο για την Επιτροπή σα να καλέσετε την μελλοντική διευθύντρια. Ε, και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σα λόγια. όταν μιλάμε για 4.000 και για 800 τετραγωνικά μέτρα, προφανώ το μουσείο δεν είναι πολύ μεγάλο. Όμω δεν είναι και ασήμαντο ω μέγεθο. θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η παρουσίαση στην μόνιμη έκθεση θα πρέπει να είναι ε, ουδέτερη από πολιτικής πλευράς. Ε, ε, να μην είναι κομματικοποιημένη. Βέβαια, το κοινοβούλιο είναι το πιο πολιτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και γι' αυτό το λόγο ίσως οι προσωρινές εκθέσεις θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες. Θα μπορούσαν να καταλάβω, να κατανοήσω ότι ε, οι άνθρωποι που ανήκουν στη δική μου πολιτική οικογένεια θα ενδεχομένως θα ήθελαν να δουν μια έκθεση για την ε, εξέλιξη της συμμετοχής των γυναικών στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να ζητήσουν μια έκθεση για την χριστιανοσύνη στην Ευρώπη κλπ ή κάποιοι άλλοι για την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα ανά τους αιώνες. Ε, εκεί στις προσωρινές εκθέσεις θα μπορούσαμε ε, όχι μόνο να προάγουμε την πολυφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και να ε, φιλοξενούμε εκθέσεις από αλλού, που μάλιστα μπορεί να είναι και πολύ διαφορετικές από τις δικές μας, από τη δικιά μας. το κόστος το λειτουργικό κόστος είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, ε, έτσι έχει υπολογιστεί. Και εγώ τώρα μιλάω σε εσά, έτσι είμαστε συνάδελφοι. Πόσο θα κοστίσει, ε, πόσο θα κοστίζει το 2016, δεν εξαρτάται από πολλού παράγοντε. Ο κ. Σκέλη είπε κάτι για παράδειγμα. Υποτίθεται ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν. Εκεί ε, αυτό το θέμα συζητήθηκε πολύ. Η είσοδο θα είναι δωρεάν. Δεύτερον, θα λειτουργεί έξι μέρε τη βδομάδα και μία από αυτέ τι μέρε μέχρι πολύ αργά. Οπότε, όταν ε, ε, στον υπολογισμό των δαπανών για την κατασκευή του μουσείου είμαι σίγουρος. Αλλά για τα λειτουργικά έξοδα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πόσους, θα πόσους φύλακες θα χρειαστούμε. Σε ένα κτίριο το οποίο θα λειτουργεί 18 ώρες τη μέρα. Πόσους φύλακες χρειαζόμαστε για ασφάλεια. Ειλικρινά, όταν μιλάμε για 11 ή 12 εκατομμύρια ευρώ λειτουργικό κόστος, ε, ας μην είμαστε και απόλυτοι. Ας έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το γεγονός ότι είναι, ε, δεν είναι ένα απόλυτο νούμερο. Είναι κατά προσέγγιση. Ο κύριος Τόκες, ε, η συνεισφορά ήταν πολύ σημαντική όταν ήταν πρόεδρος. Και αυτό που είπε ήταν ε, πολύ κρίσιμο. Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτό το μουσείο να αποφύγουμε τον ιστορικό μανιχαϊσμό στην σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης ε, έχουμε πάντοτε ε, τους καλούς, τους δυτικούς κατά παράδοση και τους κακούς που ήταν οι Ανατολικοί. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εγώ ήμουν στη φυλακή και πολεμούσα για την ε, ελευθερία και δεν ήμουν στην Ανατολική Ευρώπη. Οπότε μετά τον ψυχρό πόλεμο μάλλον κατά τη διάρκεια του ε, ψυχρού πολέμου είχαμε δικτατορίες που καταπίεζαν τους λαούς και εδώ και εκεί. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε και να υπογραμμίσουμε και την αλληλεγγύη των μεν και των δε που πάλευαν και αγωνιζόντουσαν για την ελευθερία και τα δικαιώματα όλων. Και να θα θυμόμαστε ότι υπήρχαν και κάποιοι οποίοι υποστήριζαν αυτούς που μαχόντουσαν. Γιατί και αυτό έχει σχέση με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Γιατί και στις δύο μεριέ υπήρχαν υποστηρικτές αυτών που πάλευαν για τι ελευθερίε στην άλλη μεριά. Στην Ουγγαρία το 1956, στην Τσεχοσλοβακία το 1967, ε, η υποστήριξη των ε, Ισπανών μαχητών του Οφιλίου Πολέμου, ε, των Δημοκρατικών, όλα αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και η αλληλεγγύη εκφραζόταν από ανθρώπους που δεν είχαν ενδεχομένω επισκεφθεί ποτέ τη χώρα μου ή τη δική σας χώρα. Γιατί και την υποστήριζαν ε, την, τους αγώνες αυτούς γιατί οι αγώνες αυτοί αποτελούσαν ελπίδα. Τώρα, μειονότητες και θρησκείες. Ασφαλώς και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι θρησκείες είναι κάτι πολύ δύσκολο όμως. Θα το κάνουμε όμως με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να δούμε την επίδραση της ιστορίας στη θρησκεία. Η χώρα μου για 800 χρόνια ήταν μουσουλμανική χώρα. Δεν ήταν μια χώρα η οποία έγινε μουσουλμανική λόγω εισβολής. 10.000 ήταν αυτοί οι οποίοι ήρθαν στην Ισπανία από τις αραβικές περιοχές. Αλλά για 800 χρόνια είχαμε ανθρώπους που γεννιόζησαν στην Ισπανία σαν μουσουλμάνοι. Στις περιοχές που ήταν κάτω από μουσουλμανική, μουσουλμανικό έλεγχο. Αλλά εκεί υπήρχε ανεξιθρησκεία και οι χριστιανοί και οι Εβραίοι μπορούσαν να ασκούν τη θρησκεία τους και υπήρξε άνθηση των τεχνών της αρχιτεκτονικής κτλ. Όταν όμως υπήρξε η ανακατάκτηση από τους χριστιανούς, οι Ιουδαίοι, οι εβραϊκές θρησκείες δεν μπορούσαν να ζήσουν εκεί και οι μουσουλμάνοι δεν μπορούσαν να ζήσουν εκεί ή έπρεπε να αλλαξοπιστήσουν ή έπρεπε να φύγουν από την περιοχή αυτή. Αυτά δεν τα λένε τα ιστορικά βιβλία. Αυτά που διδάσκουμε στα παιδιά μας που λέμε «Α, απελευθερώσαμε τη χώρα μας και διώξαμε αυτούς τους άπιστους οι οποίοι πιστεύαν σε κάτι διαφορετικό». Μα αυτοί οι άπιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι προηγουμένως είχαν τη διοίκηση αυτής της περιοχής. Είναι πολύ πολύπλοκα αυτά τα πράγματα. Σε όλες τις χώρες μας τα βιβλία, τα ιστορικά, μιλάνε για θρησκευτικούς πολέμους. Αλλά δεν είδα ποτέ να αναφέρονται οι ιστορικοί πόλεμοι, η αθλητικοί πόλεμοι, η πολιτιστικοί πόλεμοι. Οι θρησκευτικοί πόλεμοι ουσιαστικά ήταν ενδοχριστιανικη πολεμη πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι τα θρησκευτικά θέματα και τα θέματα των μειονοτήτων θα πρέπει να έχουν κάποια παρουσίαση σε αυτό το μουσείο. Και εδώ έχουμε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, γιατί αυτό το εγχείρημα είναι ένα σατανικά δύσκολο. Το λέω αυτό ως άθεος, ως μη χριστιανός. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Η κυρία Βερζιά νομίζω ότι απήντησα αυτά τα οποία αναφέρατε. Πράγματι δεν μπορεί να αναφέρεται μονάχα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε από 6 χώρες και έχει φτάσει στις 27 και σε λίγο 28. Και κάποια από αυτά τα κράτη, όπως η Κροατία, δεν ήταν καν ανεξάρτητα κράτη όταν ξεκίνησε το γίγνεσθε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά και δείχνει το πόσο σημαντικό είναι. Μέσω αυτών που θα δείξουμε σε αυτό το μουσείο θα μπορέσουν οι επισκέπτες να δούνε με ένα πιο πολύπλευρο πρίσμα τα προβλήματα της Ευρώπης και θα ξεπεράσουν τη μονομερή αντιμετώπιση που είδανε και μόνο στα σχολικά βιβλία. Κύριε Σκούρια, όταν λαμβάνετε το λόγο, συγκινούμε από αυτά που λέτε. Είσαστε από τα άτομα τα οποία γεννούν βαθιά αισθήματα σε μένα. Καταλαβαίνω κι εγώ αυτό που λέτε, πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση. Όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ αυτό το εγχείρημα μαζί με τον κύριο Πέτριν, δεν θεωρούσα ποτέ ότι θα φτάσουμε σε ένα πέρας, ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε, αλλά σε κάτι θετικό. Θεώρησα όμως ότι έπρεπε να το προσπαθήσουμε, αλλά ήταν τόσο δύσκολο για μένα που στην αρχή δεν θεωρούσα ότι θα ευδοκιμούσε αυτό το εγχείρημα. Γιατί για να συνενώσει κανείς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ξεπεράσουμε την, ε, τις προκλήσεις αυτές είναι πολύ δύσκολο. Η Γερμανία έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα φαντάσματα του παρελθόντος. Άλλες χώρες όμως δεν το έχουν πετύχει αυτό ακόμα. Υπάρχουν πολλέ χώρες οι οποίοι προσπαθούν επί χρόνια να φτάσουν σε κάτι αντίστοιχο και το σχέδιο αυτό είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από 20 χρόνια. Έχει αποτύχει στο παρελθόν. Κάθε φορά ήταν πάρα πολύ μάγειροι στην κουζίνα και παίζανε ξύλο μεταξύ του. Ενώ τώρα υπάρχει ένα κοινοβούλιο το οποίο μπορεί να προωθήσει με ενιαία αντιμετώπιση αυτή την ιδέα. Ελπίζω λοιπόν θα επιτύχει αυτό το εγχείρημα. Ο κύριος Στάκουλα, α, ο κύριος Στάκουλα δεν είναι πια εδώ. Δεν χρειάζεται να το απαντήσω, αλλά θα ήθελα να πω και σε αυτόν και στον κύριο Κέλλη. Ο χριστιανισμός, φυσικά, ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι ο χριστιανισμός είναι ένα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ε, αυτό όμως δεν σημαίνει είναι ότι είναι το κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι. Υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην ευρωπαϊκή ιστορία. Και νομίζω ότι και ο κύριος Σκούρια έχει τονίσει πολύ σωστά ότι υπάρχουν πολλές πολιτιστικές ιδίω τάσεις οι οποίες στεγνώριζαν σύνορα. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε πόσο εύκολα μπορούσε να περάσει κανείς από ένα μέρος στην Ευρώπη χωρίς διαβατήριο αυτοί οι οποίοι είχαν γεννηθεί παραγωγικά στην ε, Τρανσιλβανία ήταν τμήματα της αυστρο Αυτοκρατορίας ήταν νέοι με μια συγκεκριμένη πικότητα και μετά άλλαξαν πάλι πικότητα, άλλαξαν εθνικότητα. Ήταν μια γυραιά κυρία η οποία ήταν βιολονίστρια και μου έλεγε πως πήγαινε από την Τρασιλβανία στην Άγια Πετρούπολη. Αυτά γινόντουσαν στο 10ο ένα το αιώνα. Και έλεγα πώς το κάνατε αυτό, τι είχατε, είχατε κορώνες, τι δυνάρια, τι είδους νομίσματα είχατε, τι παίζατε, τι είδους μουσική. Δεν υπήρχε λοιπόν η αντιμετώπιση του ότι κάποιο θα συμβρανώσει, είναι Εβραίο ή οτιδήποτε. Δεν είχε καμία σημασία τότε. υπήρχαν Ούγγροι οι οποίοι μιλούσαν σλοβακικά. <clears throat> Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα εκείνη την εποχή. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Κέλλη. Αυτό το οποίο παραμένει σημαντικό είναι ότι αυτό το εγχείρημα είχε καταρχήν πάρα πολλούς αντίπαλους, εχθρούς σε αυτό το σχέδιο. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι αντιευρωπαϊστές κατά της ευρωπαϊκής οικοδόμησης ήταν αντίπαλοι αυτού του σχεδίου. Υπήρχαν όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε «Μα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ταυτότητα, δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή ιστορία». Μα μου πει κάποιος ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ιστορία, πώς θα τον πεις ότι θέλει να έχει ένα μουσείο Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, Ήταν, Ευρωπαϊκή Ιστορία ήταν πολύ τέτοιοι. Και ήταν και οι άλλοι οι οποίοι είπαν γιατί το κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι μια λογική ιδέα. Γιατί δεν έχει ποτέ εμπλακεί ένα κοινοβούλιο στη δημιουργία ενό τέτοιου οίκου ιστορία. Αλλά η απάντηση ήταν να το κάνουμε εμεί, να το κάνει κανεί. Και είναι κάτι που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Χρειάζεται να δείξουμε στους ε, πολίτες της Ευρώπης ποια είναι η ταυτότητα της Ευρώπης και πώς πετύχαμε να φτάσουμε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Άλλοι λέγανε ότι καλό είναι αυτό το εγχείρημα, αλλά έχουμε τώρα οικονομική κρίση. Με οικονομική κρίση δεν μπορούμε να δαπανίσουμε χρήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό είναι, ένα, είναι κάτι, ένα ρεφρέν που ακούω πάντα με τη, τα πολιτιστικά θέματα, ότι δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα τα πολιτιστικά θέματα μου. Χρειάστηκε να πείσουμε πάρα πολλούς και καταφέραμε να πείσουμε πολλούς από αυτούς. Παραμένουν βέβαια πολλοί σκεπτικιστές και ιδίως στις βρετανικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας όπου εκεί έχουν μεγάλη επιρροή ακόμα και σε ευρωπαϊστικές χώρες όπως η Γερμανία υπάρχουν ερωτήματα πρέπει να προχωρήσουμε ή όχι μήπως είναι χαμένος χρόνος, χαμένο εγχείρημα, μήπως πετάμε λεφτά. Νομίζω ότι αυτά είναι λογικά επιχειρήματα και εκεί πρέπει να εξηγήσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Και τέλος για τον κύριο Μπόρις, θέλω να επιμείνω. Δυστυχώς υπάρχουν διοικητικές δυσκολίες, αλλά θα τις ξεπεράσουμε. Ο μόνος κίνδυνος είναι αντί να ανοίξουμε το μουσείο το 2014, να το ανοίξουμε το 2015. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, θα το ξεπεράσουμε. Και η κυρία Ντυρό, η αντιπρόεδρος κυρία Ντυρό, η οποία ήταν υπουργό στο παρελθόν στο Βέλγιο και έχει προωθήσει ενεργά το σχέδιο αυτό και έχει προωθήσει επαφές με τις βελγικές αρχές. Έχουμε ξεπεράσει το οικονομικό θέμα αλλά αυτό που δεν πρέπει να επιτρέψουμε είναι να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο προπολογισμό του σχεδίου, γιατί αυτό θα είναι πολύ επικίνδυνο. Και τέλος, πρέπει να κατανοήσουμε και δύο συμπληρωματικότητες. Καταρχήν, θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα η μόνιμη έκθεση και οι προσωρινές εκθέσεις και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, του Παρλαμεντάριου και της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έλεγα. Και επιπλέον δεν θα δείχνει την αρχαία ιστορία της Ευρώπης το μουσείο αυτό. Καταλαβαίνω πρέπει να υπάρχει κάτι που να λέμε για τον Μεσαίωνα κτλ. Αλλά είναι μουσείο σύγχρονης ιστορίας. Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να πω ότι είναι δύσκολο για μας να κάνουμε κατανοητό ότι αυτό το σχέδιο είναι όχι μόνο χρήσιμο αλλά και απαραίτητο. Για κάποιους από εμά, όχι ίσως για σας, αλλά για αυτούς οι οποίοι έρχονται από τη δική μου γενιά <clears throat> και για αυτούς που είναι λίγο μικρότεροι από μένα αλλά κοντά στη γενιά μου όπως είναι η Ντόρις, αυτό το μουσείο θα είναι συγκινητικό γιατί είναι ουσιαστικά η ιστόρηση της δικής μας ζωής και πορείας. έχω πει ότι το μουσείο αυτό δεν πρέπει να είναι για μας, για τη γενιά μας, να είναι ένας καθρέφτης όπου ξαναβλέπουμε τον εαυτό μας. Η πρόκληση είναι αυτό το μουσείο να μιλάει και στα παιδιά μας, σε αυτούς που δεν έχουν ζήσει τη δική μας εποχή και για τα παιδιά των παιδιών μας, που δεν έχουν καμία ιδέα για όλα αυτά τα γεγονότα. Στη χώρα μου εγώ με πολλές φορές όταν βλέπω ότι παιδιά 10 ετών λένε ότι ο στρατηγός Φράνκο και οι καθολικοί ε, βασιλιάδες που ήταν στο 15ο αιώνα ο... βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή 50 χρόνια πριν από 50 χρόνια και 500 χρόνια πριν για ένα παιδί 10 χρόνων είναι το ίδιο πράγμα. Έχει συμπυκνωθεί η ιστορία. Είναι ένα ορίζον και δεν βλέπουν ότι η μια εποχή είναι διαφορετική εποχή, ότι έχουν περάσει 450 χρόνια ανάμεσα. Η πραγματική πρόκληση λοιπόν είναι να μην φτιάξουμε κάτι το οποίο θα προβάλλει τη δική μας εμπειρία, αλλά να είμαστε αρκετά γενναιόδοροι για να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα μιλάει στα παιδιά μας και τα αγκόνια μας. Σας ευχαριστώ πάλι και για την προσοχή σας και ελπίζω ότι θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε και με τη Διευθύντρια του Μουσείου. Ωραία. Υπάρχουν τα χειροκροτήματα αυτά, τα οποία τα έχει κερδίσει πράγματι ο κύριος ε, Ματίνες, γιατί χρειάζεται και μία συγκινησιακή προσέγγιση στα θέματα αυτά. Ο κύριος Ματίνες και ο κύριος Πέτερινγκ έχουν προωθήσει αυτό το σχέδιο και βλέπετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχείρημα. Αν δεν προχωρήσουμε και το έκανε κάποιο άλλο, δεν θα είχαμε καμιά δυνατότητα επιρροή. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό ο οίκο τη Ευρώπη και με το πνεύμα που σας περιέγραψε ο κύριος Μαρτένη, ελπίζω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα την ευκαιρία να μιλήσουμε με τη διευθύντρια του μουσείου. Δεν θέλησε τώρα να παρέμβει και να ε, παρεμποδίσει την έκφραση των απόψεών μας, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτό το σχέδιο και θέλω να σε ευχαριστήσω αγαπητέ ε, Άγγελ και συνεχίζουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημέρησης διάταξης. Μέρση αμπιεντό. Ok. Bon, alors, ça fait du bien, hein <laughs> Bon, ok. Euh, we have only, only one, um, one uh, point of the agenda. Ένα σημείο ακόμα στην ημέρησια διάταξη έχουμε και το απόγευμα θα έχουμε τον ε, Γενικό Διευθυντή που θα μας επισκεφτεί. Έχουμε τώρα το σημείο που αφορά που έχει να κάνει με την πρόθεση εθελοντικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 20 Σεπτεμβρίου πέρσι η Κομισιόν δημοσίευσε μια ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Εθελοντισμό και φυσικά πέστανε το έτος του εθελοντισμού η ανακοίνωση αυτή που είχε να κάνει με την αναγνώριση και την πρόθεση των διαμεθοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να ακούσουμε από τον κύριο Σκουρία ποια είναι η άποψή του για αυτή την ανακοίνωση και πώς την κρίνει. Σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο και μετά από αυτή τη συζήτηση έχουμε τη συνάντηση, τη συνεδρίαση των συντονιστών μετά γίνεται τη διακοπή και επανερχόμαστε το απόγευμα. Κύριε Σκουρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο το δυνατόν λιγότερο ώστε να δώσουμε το λόγο και στους συναδέλφους. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Φοντανίνη από τη Γραμματεία με την οποία συνεργάστηκα εξαιρετικά και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους οποίους ε, συναντηθήκαμε προκειμένου να εμβαθύνουμε κάποιες πτυχές του συγκεκριμένου ζητήματος. Ευθύ εξ αρχή ε, θεωρήσαμε ότι δύο σημεία είναι σημαντικά. Καταρχά θα πρέπει να ε, τελειοποιήσουμε τον ορισμό του εθελοντισμού διότι ξέρουμε ότι δημιουργεί ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στα κράτη-μέλη κάποιες ε, διαφορές στην ερμηνεία και θελήσαμε να επισημάνουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο εθελοντισμό. και σε δεύτερο επίπεδο θέλαμε να επισημάνουμε και τις θετικές ε, ε, επιρροές που είχαμε από το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού το 2011, ε, διότι πέρα από τις συναντήσεις και τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών που έγιναν μεταξύ των διαφόρων συστημάτων στη διάρκεια του 2011, είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε μια χώρα, η Λιθουανία, η οποία πέρσι πέρασε τον πρώτο εθνικό νόμο για τα θέματα του εθελοντισμού. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια χρονιά η οποία δημιούργησε μια συζήτηση και προέκυψαν και κάποια αποτελέσματα. Και φυσικά πολλά κράτη-μέλη, πολλές κυβερνήσεις άρχισαν να ασχολούνται με το θέμα αυτό ξανά και ε, ε, να κάνουν έναν εξυγχρονισμό των κείμενων κανόνων σε κάποιες χώρες ε, κάτι το οποίο προέκυψε και από τη μεγάλη συζήτηση που είχαμε στη διάρκεια του 2011. Και την προηγούμενη φορά όταν ξεκίνησε η συζήτηση του θέματος αυτό είχαμε πει ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μία ανακοίνωση η οποία κατά την άποψή μας είναι καλώς καμωμένη, άρτια και Αναφέρθηκαν κάποια σημεία τα οποία θεωρήσαμε θεμελιώδους σημασίας και έχουμε προσθέσει και κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι πρέπει να την χάνει ιδιαίτερης προσοχής ο εθελοντισμός από τις αρχές υψηλού επίπεδου, ιδιαίτερα για τους λιγότερο ευνοημένους, ε, τους αναπήρους, τους ε, νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες και ούτω καθεξής. Επιπλέον έχουμε συμπεριλάβει και την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να κατανοήσουν και να γνωρίζουν τι δυνατότητες προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη για θέματα εθελοντισμού και συζητήθηκε η δυνατότητα να υπάρχει μια κεντρική δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει και συγκεκριμένο τμήμα αφιερωμένο στον εθελοντισμό που θα εξηγεί προγράμματα, δυνατότητες, ε, κόστος και ευκαιρίες για όσους θέλουν να συμμετέχουν. Θελήσαμε επίσης να επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να έχουν ε, μία μέθοδο μέτρησης των αποτελεσμάτων του εθελοντισμού, ε, τα οποία στοιχεία γνωρίσαμε σε κάποιες συναντήσεις. Ε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο John Hopkins και έχει υιοθετήσει και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας για να υπάρχει ένα στοιχείο μέτρησης ε, ε, και σύγκρισης ε, των θεμάτων εθελοντισμού, κάτι το οποίο δεν υπάρχει τη σήμερον ημέρα και γιατί είναι πολύ διαφορετική η νομοθεσία και τα μέσα τα οποία υπάρχουν και πολλές φορές είναι δύσκολο να εξετάσουμε τα θέματα αυτά εις βάθος. Βεβαίως αναφέρθηκε στη διάρκεια του έτους αυτού και το έτος ενεργού γύρανσης, ε, το πόσο σημαντική είναι ε, η εθελοντική εργασία για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Αναφέρθηκε επίσης πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός, ε, διότι υπάρχει και νέα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό και υπάρχει και μια έκθεση που εγκρίναμε πριν από κάποιους μήνες εδώ στην Επιτροπή μας και στη συνέχεια στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για τη σημασία του αθλητισμού και τη σημασία του εθελοντισμού στον αθλητισμό. Επισημαίνεται επίσης και καλούνται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν τη δέουσα σημασία στον εθελοντισμό ε, και το πώς ε, ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των εδαφών, ε, την πολιτιστική κληρονομιά, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές φυσικές και περιβαλλοντικές καταστροφές που πλήττουν την Ευρώπη και ίσως θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση από αυτού. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός εθελοντικού ανθρωπιστικού σώματος είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όπως επίσης και η πρόταση του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Δεξιοτήτων, ώστε όλες οι δεξιότητες που αποκτούνται μέσω του εθελοντισμού να αναγνωρίζονται επισήμως ε, και από επαγγελματική σκοπιά, αλλά και ε, με στόχο να μαθαίνει κάποιος περισσότερο και να ε, συμπληρώνεται το βιογραφικό των εθελοντών με δεξιότητες οι οποίες έχουν αποκτήσει μέσω του εθελοντισμού. Επισημάναμε επίσης πόσο σημαντικές είναι οι διάφορες οργανώσεις και πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στον τομέα αυτό. Χωρί αυτέ τι οργανώσει φυσικά δεν θα μπορούσε καν να αναφέρεται ο όρο εθελοντισμό και επομένω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν περαιτέρω μέσα ε, χρηματοοικονομική βοήθεια και στήριξη, ιδιαίτερα τώρα σε καιρού κρίση, διότι σε αυτέ τι στιγμέ ο εθελοντισμό είναι αυτό ο οποίο δίνει απαντήσει και ορισμένε φορέ αποτελεί υποκατάστατο ε, των τοπικών και κρατικών αρχών όταν δεν μπορούν να παρέμβουν απευθεία. Κάτι που μας άρεσε επίσης ήταν το γεγονός ότι αναφέρουμε στις αιτιολογικές σκέψεις ότι ο θελοντισμός αποτελεί στοιχείο διαλόγου με τον υπόλοιπο κόσμο, με όλες τις χώρες δηλαδή οι οποίες δεν είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα και μέσω του εθελοντισμού μπορούμε με κάποια περηφάνεια να ε, παρουσιάσουμε το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική συνοχή, δύο πτυχές τις οποίες θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές για τις κοινωνίες μας και όχι μόνον. Αυτά λοιπόν εν συντομία. Υπάρχει βέβαια και η έκθεση την οποία μπορείτε να διαβάσετε όλοι και να παρουσιάσετε και τροπολογίες. Αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και φυσικά είμαι εν αναμονή των παρατηρήσεών σας ε, για να διαμορφωθεί στη συνέχεια η έκθεση, ε, μια έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει ε, όλα τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω ότι ο εισηγητής γνωρίζει πολύ καλά το χώρο του εθελοντισμού και η έκθεση αυτή είναι πολύ καλά συντεταγμένη. Μπορεί να υπάρξουν μικρές βελτιώσεις, αλλά συμφωνώ με την κύρια γραμμή που ακολουθεί ο εισηγητής και χαίρομαι για το γεγονός ότι τονίζει την ανάγκη, στην αρχή την ανάγκη να υπάρχει μια καθαρή γραμμή για τα θέματα των ε, εθελοντών. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο το οποίο θα δημιουργηθεί το οποίο θα επιτρέψει η δραστηριότητα των ε, εθελοντών να λειτουργήσει σωστά. Χαίρομαι που η Σλοβακία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που ενέκρινε νομοθεσία για τους εθελοντές. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να βασιστούμε σε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Για το τρίτο σημείο τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει εμείς να τονίσουμε ότι θέλουμε να υπάρξει και ο εθελοντισμός για τους Ρώμα. Ας διευρύνουμε για να μιλήσουμε για όλες τις μειονοτικές ομάδες. Το να μιλάμε μονάχα για τους Ρώμα <clears throat> δεν είναι ίσως τόσο θετικό. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Στο σημείο 7 επίσης ο εισηγητής ζητά να υπάρχει μια δικτυακή πύλη για την, τον εθελοντισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν υποστηρίζω τη δημιουργία νέων πυλών, νέων γραμμών του προϋπολογισμού, νέων ε, φορέων. Ίσως μπορούν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης να βρουν από τα κράτη-μέλη τους την, ε, τις πληροφορίες που θέλουν για το πώς να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές ενέργειες. αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πάνω από 100 εκατομμύρια πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε κάποιο βαθμό εθελοντές και ίσως μπορούμε να ευξήσουμε αυτόν τον αριθμό. Επίσης πρέπει να ξέρουμε πώς θα καταμετρούμε τη δραστηριότητα των εθελοντών. Δεν είναι μονάχα ένα θέμα της ε, αξίας τους ή της αμοιβή τους από την ε, κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχει όμως ένας τρόπος ποσοτικοποίησης της έντασης εθελοντισμού. Όπως όταν υπολογίζουμε μια σύνταξη, θα πρέπει κάπου ο εθελοντισμός που δεν είναι αμοιβόμενη εργασία να υπολογίζεται και για τον για τη σύνταξη που παίρνει ένα άτομο. Επίσης θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λαμβάνουμε υπόψη την άτυπη παιδεία και τις δεξιότητες που αποκτά κανείς με τον εθελοντισμό. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει κάπου να την χάνουν και κάποιες αναγνώσεις. Πολύ σωστά τα λέει ο στο σημείο 12. Σημείο 14. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών για ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα είχαμε και περισσότερους εθελοντές οι οποίοι θα μπορούν να, ε, να συνδράμουν σε ανθρωπιστικές καταστροφές και αυτό θα βοηθούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να, δίνει, να έχει μια καλύτερη εικόνα προς τον εξωκόσμο και να είναι παρούσα εκεί που υπάρχει ανάγκη. Κάτι το οποίο λείπει και το οποίο θα προτείνω σαν ανθρωπολογία είναι το πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εθελοντές. Χρειάζεται να τους δώσουμε περισσότερες δυνατότητες, να έχουν περισσότερα περισσότερε δυνατότητε στέγαση εκεί που χρειαζόμαστε εθελοντές και μια άλλη πτυχή. Ο εθελοντισμό δεν αφορά μόνο τους Ευρωπαίους, αφορά όλους του ανθρώπους στον πλανήτη μας. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτού που ζουν εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαμε ίσως να <clears throat> δημιουργήσουμε ένα μοντέλο που θα δίνει και πιο μεγάλη ευκολία <clears throat> με πιο μεγάλη ευκολία να δίνει προξενικές θεωρήσεις σε αυτούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν σε εθελοντικές δραστηριότητε και έτσι να διευκολύνουμε τη συμμετοχή του σε τέτοιε ενέργειε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάω μόνο για ανθρωπιστικέ καταστροφέ, αλλά μιλάω και για νέου οι οποίοι έρχονται ω εθελοντέ στην Ευρώπη και θα βοηθήσουν ενεργά χώρου που υπάρχουν προβλήματα και ανάγκε. Και φυσικά μιλάμε κυρίω για νέου και εν κατακλείδη εγώ σύμφωνο με αυτά τα οποία λέει ο εισηγητής ότι πρέπει να δώσουμε και μια οικονομική ενίσχυση στις εθελοντικές δραστηριότητες και να συμπεριληφθούν στις μελλοντικέ δαπάνες στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν μονάχα αν έχουν την <clears throat> χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς θα πρέπει να δίνουμε χορηγίες σε αυτές τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Θέλω να παρακαλέσω τους επόμενους ομιλητές να είναι κάπως πιο σύντομοι, γιατί έχουμε και τη συνάντηση των συντονιστών στη συνέχεια και δεν θα έχουμε διερμηνία άμα δεν τελειώσουμε εγκαίρως. Η κυρία Σάνσεθ Σμιτ έχει το λόγο. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουριά, το, ο οποίος εξέτασε πολύ πλευρά το θέμα. Έχει πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα που μας επιτρέπουν την μέτρηση της σημασίας ε, του εθελοντισμού. Θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη που ανέφερε να γίνει μια απογραφή, μια σαφής απογραφή για να αξιοποιήσουμε και να προβάλλουμε τον εθελοντισμό. Υπάρχουν μέσα που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα στους εθελοντές και στις ενώσεις τους προκειμένου να αναπτυχθούν και προκειμένου να τους εξυπηρετήσουν στις δραστηριότητε τους. Για παράδειγμα, ε, υπάρχουσες ρυθμίσεις για την διασυνορική συνεργασία, στόχος 3 της πολιτικής συνοχής. Αυτές οι διατάξεις ε, θα πρέπει να είναι γνωστές από τους εθελοντές, θα πρέπει να τους γίνουν γνωστές, συνεπώς ε, θα ε, πρέπει να προωθήσουμε την εικόνα των ε, ευρωπαϊκών ε, ταμείων ενώπιον των εθελοντών και να προωθήσουμε και την χρήση περιφερειακών ταμείων για διασυνοριακά προγράμματα εθελοντισμού. Σύμφωνα με τους στόχους που έχουμε, η συμμετοχή των πολιτών, ενεργή γύρανση, νεότητα, τα ε, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή κλπ. Όλοι αυτοί οι στόχοι της κοινωνικής συνοχής ε, στην εδαφική συνεργασία ε, προβλέπουν δράσεις όπως δημιουργία δικτύων, ανταλλαγή καλών βέλτιστων πρακτικών κλπ. Και μην ξεχνάμε ότι μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από τον άλλο. Για παράδειγμα, ο νόμος 1901 της Γαλλίας για τις ενώσει εθελοντών. Ευχαριστώ την κυρία Σάντσε Σμιθ. Ο κύριος Έρβαρτ τώρα έχει το λόγο. Thank θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το άρτιο έργο του στο θέμα αυτό. Υποστηρίζω τα όσα αναφέρει η έκθεση για καλύτερη ο συντονισμό των εθελοντικών δραστηριοτήτων και την προαγωγή της κινητικότητας ε, των εθελοντών ανά την Ευρώπη. Αυτό ε, το θέμα επίσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Δικτυακής Πύλης ε, θα δημιουργήσει τη δυνατότητα να συντονίζονται καλύτερα ε, οι εθελοντές. Οι διάφοροι οργανισμοί και οι λέσχες ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι ακριβώς τους προσφέρεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η γραφειοκρατία για την χρηματοδότηση ορισμένες φορές αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Καλό είναι λοιπόν να εφαρμόζονται διαμεθοριακά κριτήρια και δυστυχώς επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν αυτά τα κριτήρια, κάποια πολύ καλά προγράμματα και ιδέες δεν προχωρούν. Δεν μπορεί κάποιος να προχωρήσει τις ιδέες του στο επόμενο ε, στάδιο. Μια κεντρική λοιπόν δικτυακή πύλη η οποία θα μπορεί να προσφέρει υποστήριξη και να δημιουργήσει ένα δίκτυο σίγουρα θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα που θα ενισχύσει το ρόλο και τη συνεισφορά των οργανώσεων εθελοντών και θα μπορέσει να δημιουργήσει συμμετοχικές κοινωνίες. Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων θα ενισχύσει σημαντικό το ρόλο των εθελοντών και θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε και την κινητικότητά τους. Η σημαντική συνεισφορά αυτού του διαβατηρίου θα πρέπει ίσως να αναφερθεί λίγο περισσότερο στην έκθεση, διότι θα δώσει κίνητρα στους εθελοντές και θα αυξήσει και την ε, συμμετοχή. η σημασία του εθελοντισμού στον αθλητισμό, στην έκθεση που είχαμε για τον εθελοντισμό, ήταν πολύ σημαντική. Υπήρχαν κάποιε πρωτοβουλίε, τι οποίε καλό θα ήταν ίσω να αναφέρουμε και στην έκθεση αυτή. Το γεγονό ότι 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε συμμετέχουν σε κάποια μορφή εθελοντική προσφορά είναι σημαντικό στοιχείο και θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση για να υποστηρίξουμε τι οργανώσει εθελοντών. Χωρίς μικρόφωνο Δίνει τώρα στην κυρία και εγώ μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ευχαριστώ τον Μάρκο Σκούρια. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό έδαφος για την περαιτέρω συζήτηση. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι ε, είδους αιτήσει θα πρέπει να διατυπώσουμε προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη, θα είναι χρήσιμο να κάνουμε να διτυπώσουμε και εκκλήσεις προς τις επιχειρήσεις στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο να αναγνωρίζουν δηλαδή, την εθελοντική δραστηριότητα των εργαζομένων της, αλλά να την υποστηρίζουν ενεργά όταν είναι εθελοντές οι εργαζόμενοι. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια υπάρχει η επιχείρηση Henkel, η οποία έχει όχι μόνο υποστήριξη προς τους εργαζομένους αλλά και η ίδια βοηθά και προωθεί τους ε, εργαζομένους της σε τέτοιες ενέργειες τις οποίες διενεργεί και η ίδια η εταιρεία. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια έκκληση προς τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αυτό θα μπορούσε να είναι θετικό στοιχείο πρόσθετο σε αυτά που αναφέρει ο συγητής. Κύριος Μάτουλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα. Αν ξεκινήσουμε από τον βασικό ρόλο που έχει η... ο εθελοντισμός και τα πορίσματα του ευρωπαϊκού έτους για τον εθελοντισμό, μπορούμε να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή, ο εθελοντισμός αναπτύσσεται όλο και περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί είναι όλο και πιο σημαντικά. Δυστυχώς όμως τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα νομικά, νομοθετικά εμπόδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένουν πολλές φορές ανυπέρβλητα και ακυρώνουν ένα τμήμα των θετικών αποτελεσμάτων του εθελοντισμού. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι και να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά. Αν θέλουμε εμείς να αρχίσουμε να ελέγχουμε το διαδίκτυο σε ευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να ζητήσουμε από τα ευρωπαϊκά κράτη όχι μόνο να έχουν μια σαφή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα θέματα του εθελοντισμού, αλλά και από την Κομισιόν να κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι σε αυτή τη χρονική στιγμή να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερούμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε στο μέλλον μια δραστηριότητα που είναι τόσο σημαντική, τόσο χρήσιμη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλω να συγχαρώ τον ε, συνάδελφό μας, τον κύριο Σκουρία. Το έγγραφο εργασίας είναι πολύ πραγματιστικό, πολύ χρήσιμο. Εγώ θα το υποστηρίξω και η ελπίση μου είναι ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάρκο, θες να πεις κάτι εν Α, συγγνώμη. Η κυρία Βέζια. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Θα προχωρήσω να προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί έχω και μια άλλη συνεδρία. Συγγνώμη κύριε Σκουρία, δεν έχω διαβάσει απόλυτα ακόμα την, την έκθεσή σας. Αλλά σίγουρα μετά από αυτά που έχω ακούσει υποστηρίζω ιδιαίτερα τις γενικές γραμμές της παρουσίασής σας, της πρότασής σας. Στέκομαι μονάχα σε δύο ή τρία πράγματα. Εγώ εξετίμησα ιδιαίτερα την ε, παράγραφο 17, την Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτών. Για μένα είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε ότι ο εθελοντισμός είναι και ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ε, πραγματική ενεργή συμμετοχή των πολιτών από τότε που αποκεφαλίσαμε τον τελευταίο βασιλιά στην, ε, στη Γαλλία έχουμε πάντα μια αντιπαράθεση μεταξύ της έννοιας του πολίτη και του υπηκόου. Αυτό παρενθετικά. Πάντως μέσα από αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς δια μεθοριακού εθελοντισμού στην Ευρώπη. Εξακολουθώ να τρέφω ακόμα μια γαλλογε... γαλλογαλλική επιφύλαξη. Δεν νομίζω ότι στα γαλλικά ο εθελοντισμός να αναφέρεται ως βολονταριά στα γαλλικά. Στα γαλλικά λέγεται μπενεβολά και όχι βολονταριά. Δεν θέλουμε αυτό τον αγγλοβαρβαρισμό του βολονταριά, γιατί στη Γαλλία οδηγεί σε σύγχυση στον εγκέφαλο των πολιτών. Γι' αυτό θα κάνω και γλωσσικές τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Και επίσης νομίζω πρέπει να δώσουμε και κάποια μηνύματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις των πολιτών όταν εργάζονται δημοκρατικά, που γίνεται τις περισσότερες φορές αλλά όχι πάντα, να έχουμε ένα μήνυμα να υπάρχει δημοκρατική λειτουργία των εθελοντικών οργανισμών και να τονίσουμε επίσης και την ανάγκη να υπάρχει πλήρης πρόσβαση των γυναικών στους φορείς αυτούς και στις διευθύνουσε δομέ του. Νομίζω λοιπόν ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις μειονότητε και στην εκπροσώπηση των μειονοτήτων σε αυτό το τομέα. Φυσικά υπάρχει ποικιλία καταστάσεων από ένα κράτο μέρο σε άλλο και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Κυρία Βερσιά, είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσετε να βρείτε τη σωστή έκφραση για το γαλλικό κείμενο. Αν δεν σας αρέσει το βολοντάρια, αν υπάρχει μια τέτοια διατύπωση λοιπόν, εσείς πρέπει να κάνετε και μια ε, υπόδειξη στους μεταφραστές για να τονίσετε ότι η σωστή λέξη είναι περιβολά, και όχι βολοντάρια. Μπορείτε λοιπόν να υποστηρίξετε τα γαλλικά συμφέροντα εναντί των μεταφραστών. Μάρκο, θε να πει κάτι ακόμα. Ε, Απλώ ε, να πω ότι θα συζητήσουμε και με τους κοιόδης εισηγητές ε, για να δούμε κάποια πράγματα τα οποία επισημαίνουμε. Για τον εθελοντισμό έχουμε γράψει επακριβώς τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο εθελοντισμό, ώστε πέρα από κάθε γλώσσα να είναι σαφές στους πολίτες μας σε τι αναφερόμαστε ε, Βεβαίω, από εκεί και πέρα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποιε προτάσει των ε, συναδέλφων. Τους ευχαριστώ όλους ε, για όσα είπαν εδώ, τι μειονότητε, το να γνωρίζουμε σε τι βαθμό είναι ο εθελοντισμό, της επιχειρήσει και την αναγνώρισή τους. Αυτά θα τα δούμε και με του κοιόδη ηγητές. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους. Κλείνω λοιπόν τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ όλου του παρόντε και οι οποίοι έχουν συμβάλει να γίνει η Ευρώπη πιο φιλική προς τους ε, νέους. Α, προθεσμίες. 9 Μαρτίου. 9 Μαρτίου το μεσημέρι. High noon. Εντάξει. Καλή όρεξη και οι συντονιστές μένουν στην αίθουσα. Et ceux qui sont invités.